Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, σήμερα το πρωί. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να καλοχαιρετήσω, να υποδεχθούμε την Ουγγρική Προεδρία. Σε αυτή την περίπτωση τον κύριο Υπουργό Τάμας Βέλετη, ε, που είναι Υπουργό Εθνικών Πόρων και Ανάπτυξης της Ουγγαρίας ε, και τον κύριο Υπουργό... Πέτερ Λάιος και όλη την ομάδα τους. Καλώς ήρθατε. είδαμε ήδη την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Περιβάλλοντος στην Γκέντ. Τους είχαμε ξαναδεί και θα ξανασυναντηθούμε στην παρόμοια αυτή σύνθεση στο, στη συνάντηση στην Ουγγαρία. Ο Υπουργός Ελέτη είναι αρμόδιος για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα θέμα που ιδιαίτερα στην Ευρωβουλή και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει υψηλή προτεραιότητα. Εργαστήκαμε ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος υπό τις πιο διαφορετικές πολυσχηδείς πτυχές και στο Κανκούν επίσης είχαμε ένα αποτέλεσμα που σφαιρικά, συνολικά μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας με βάση αυτό. Και κατά αυτό το εξάμεινο της Ουγγρικής Προεδρίας θέλουμε να τεθούν προτεραιότητες. Είναι ένα σημαντικό εξάμεινο, πολύ σημαντικοί έξι μήνες αυτοί όπου θα αποφασίσουμε ποια θα είναι η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός της πορείας μας. Θα συνεχίσουμε, θα είμαστε φιλόδοξοι ή θα επαναπαυθούμε στο πακέτο στη δέσμη μέτρων για το κλίμα που το 2008 αποφασίστηκε μια ολόκληρη σειρά αποφάσεων πρέπει να ρυθμιστεί και έχουμε εμπιστοσύνη και ευελπιστούμε στις προσπάθειες και την δέσμευση της Ουγγρικής κυβέρνησης υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Αλλά θα ακούσουμε από τον ίδιο. Ο ίδιος ο Υπουργός θα μας πει ποιες είναι οι δράσεις που προβλέπονται από την Προεδρία του τους επόμενους έξι μήνες. Έχει τον λόγο για την εισαγωγή στο θέμα. Στη συνέχεια αμέσως θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν συνεχίσω στα Ουγγρικά θα ήθελα πολύ σύντομα να μιλήσω στα Αγγλικά. Είναι πραγματικά τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ και να σας παρουσιάσω το κατάλογο των προτεραιοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας ε, και να σας μιλήσω σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και κυρίως στα θέματα κλιματικής αναλογής. Να σας εξηγήσω γιατί ο Υπουργός ε, ε, Επιθεμάτων Εθνικής Ανάπτυξης ασχολείται με την κλιματική αλλαγή στην Ουγγαρία. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης πριν από 7 μήνες έχουμε μια νέα δομή της κυβέρνησης και λήφθη η πολιτική απόφαση να για λόγους αποτελεσματικότητας να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες σε ένα Υπουργείο και πρόκειται για το Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης που ασχολείται με την πολιτική της συνοχής, με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιφερειακή ανάπτυξη, ενέργεια, κλίμα, ε, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και διαχείριση των κρατικών πόρων. Δηλαδή όλα όσα έχουν να κάνουν με τους πόρους και τη διαχείρισή τους ε, κυβερνητικό επίπεδο συνδέεται με το Υπουργείο μας. Ένα πολύ μικρό Υπουργείο όπως βλέπετε. Ε, θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω δύο συνεργάτες μου στα θέματα κλιματικής αλλαγής. Ο κύριος Σόλος, με ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και ο κύριος Κοάτσε είναι ε, υπεύθυνο στο Υπουργείο για τις ε, διεθνείς υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ και τώρα συνεχίζω στα Ουγγρικά. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για μας είναι πολύ σημαντικό να, να σημειωθεί πρόοδος στις διεθνεί ε, διαπραγματεύσεις για την προστασία και τι κλιματικέ ε, αλλαγέ και να έχουμε το δυνατόν πιο γοργά μια συμφωνία για την κλιματική πολιτική σε σχέση με το 2012. Είναι δυσχερή η πορεία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Για μας είναι επίση σημαντικό να έχουμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα στεφθεί με επιτυχία. Διότι όλοι θέλουμε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία που θέλουμε να αναπτυχθεί. Όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, θεωρούμε ότι η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου ανέλαβε σημαντικά βήματα και έκανε σημαντικές προόδους όσον αφορά μια φιλόδοξη, νομικά δεσμευτική συμφωνία, ένα πλαίσιο συμφωνίας ως προς αυτά η Ουγγαρία θέλει να συνεχίσει το έργο της Βελγικής Προεδρίας, όμως φυσικά θέλουμε να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες που απορρέουν από το Κανκούν. Πολλά διακυβεύονται εδώ διότι στις νοτιοαφρικανικές διαβουλεύσεις το 2011 αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία για το πώς δηλαδή η δεύτερη φάση του πρωτοκόλου του Κιώτο θα διαμορφωθεί τότε θα μπορούσε να υπάρξει ένα νομικό κενό, ένα χάσμα και αυτό θα ήταν κάτι πολύ αρνητικό θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαπραγματεύσεις και πρέπει να αποφύγουμε μια τέτοια περίπτωση. Κυρίε και κύριοι, στην διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών της ε, Συμφωνίας Πλαισίου για τις κλιματικές αλλαγές και για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το κλίμα είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα το οποίο τίθεται εδώ τις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές να τις προλάβουμε, να τις, αποφύγουμε, να τις αποφύγουμε. Αν δεν καταφέρουμε μέχρι το 2005 τις συνολικές εκπομπές ρήπων να τις μειώσουμε κατά το ίμιση σε σχέση με το επίπεδο του 1990, τότε θα έχουμε πολύ αρνητικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις παγκόσμια. Αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί σημαντικά και η πιθανότητα είναι πολύ μεγάλη να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε χώρες και περιφέρειες μπορούν να αποσταθεροποιηθούν πλήρως και θα υπάρξουν μεταναστευτικά ρεύματα από αυτές τις περιοχές προς άλλες και θα δημιουργηθεί ένα χάος. Γι' αυτό μπορεί οι κλιματικές αλλαγές να είναι πραγματικά ολέθριες και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν, να τις προλάβουμε. Τώρα, βιομηχανικές χώρες έχουν, ε, ανεπτυγμένες χώρες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις ε, όσον αφορά τις εκπομπές τρύπων. Λοιπόν, η δική μας πρόθεση είναι να είμαστε φιλόδοξοι σε σχέση με το ορόσημο 2012 και επέκεινα. Να έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο στο οποίο θα καταλήξουμε. Και αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται σε, όλους τους σημαντικούς, ε, σε όλες τις σημαντικές χώρες που εκπέμπουν ρήπους στην ατμόσφαιρα. Οι διαπραγματεύσεις στο Κανκούν σημείωσαν πρόοδους σε πολλούς τομείς σε σχέση για παράδειγμα με το 2009 και τη διάσκεψη της Κοπενχάγης του 2009. Όμως ήταν πολιτικές συμφωνίες, πολιτικές συμφωνίες αυτές ε, και για το, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του Κανκούν εμπεριέχεται επίσης ότι η μέση, ε, η οριακή τιμή αύξηση της ε, θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς ε, Κελσίου πρέπει να περιοριστεί στους 2 βαθμούς Κελσίου συνολικά. Σε ένα ψήφισμα καθορίστηκε αυτό. Επίσης ε, καθορίστηκαν υποχρεώσεις για τις αναδυόμενες χώρες και τις ανεπτυγμένες χώρες. Νέοι μηχανισμοί δημιουργήθηκαν και επίσης ε, οι μηχανισμοί για τη λειτουργία της αγοράς αξιολογήθηκαν, οι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο όργανο για να μειωθούν οι εκπομπές τρύπων μέσω εμπορίας κτλ. Στο Κανκούν καταφέραμε λοιπόν σχεδόν όλα τα σημεία να τα προσδιορίσουμε και να τα καθορίσουμε που μπορούν να αποτελέσουν τα θεμέλια για μια λειτουργική συμφωνία στο μέλλον. Στις ελλείψεις όμως ανήκει το ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για το μέλλον του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Επίσης δεν ελήφθη κάποια απόφαση για μια νέα ε, συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Και αν θα είχαμε μια συμφωνία η οποία θα ήταν υπό αυτό το πλαίσιο νομικά δεσμευτική. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα μπορούσε να, διαμορφωθεί μια τέτοια ε, συμφωνία στο μέλλον. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η υλοποίηση, η εφαρμογή της Συμφωνίας του Κανκούν. Θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της η Ουγγρική Προεδρία ώστε να μπορέσει να προετοιμάσει τις διαπραγματεύσεις του 2011. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε δύο συνεδριάσεις ε, για την ε, Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος αυτών των δύο διασκέψεων θα είναι να προετοιμαστεί η Σύνοδος Κορυφής για το κλίμα στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Επίσης η Ουγγρική Προεδρία έχει θέσει τον στόχο ενώπιόν της την θέση, την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την συντονίσει αποτελεσματικά και τις διαφορετικές τοποθετήσεις των κρατών μελών να τις προσεγγίσει αντίστοιχα ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τους εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι εξάλλου σημαντικό οι διαφορετικές θέσεις να προσεγγίσουν η μία την άλλη και να συγκεραστούν όσον αφορά το μέλλον για παράδειγμα του πρωτοκόλου του Κιώτο, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα θέματα χρηματοδότησης Επιπλέον, ένα από τα άλλα σημαντικά μας έργα, ο στόχος θα είναι οι διαπραγματεύσεις στις 12 ομάδες εργασίας να ε, συντονιστούν μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρόκειται για σημαντικές στοχοθετήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις για μειώσεις που πρέπει να επιτευχθούν, υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, ένας, έναν μηχανισμό επιπλέον ελέγχου για τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούμε και έναν μηχανισμό ευελιξίας. Όλα αυτά θα πρέπει έτσι να συντονιστούν ήδη δίνει την δυνατότητα των Κανκούν να ληφθούν συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε ε, υλοποιώντας, εκπονώντας πιο εξειδικευμένα αυτά τα μέτρα. Δημιούργησε το Κανκούν ένα νέο πλαίσιο για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει. Η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές έτσι θα διευκολυνθεί θα είναι κάτι το εφικτό και θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της αποψήλωσης των δασών και θα αντιμετωπιστεί έτσι ένα πρόβλημα με, βάση, με μια νέα βάση. Θα έχουμε μια ε, συνάντηση επαϊόντων στην Βουδαπέστη και εδώ κυρίως ε, έγινε η προσπάθεια να, καταλήξουμε σε ένα, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ε, πλαίσιο, σε μια κοινή θέση για τις διαπραγματεύσεις του 2011 στην Νότια Αφρική για το κλίμα, ξεκίνησε ανταλλαγή απόψεων για το ποια στρατηγική θα πρέπει να εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη σύνοδο για τα κλιματικά θέματα και εξετάσαμε πώς θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε η, τα μέτρα για τη Συμφωνία του Κανκούν να μπορέσουν να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Στους στόχους μας ανήκει το ότι το σύστημα MR W, το σύστημα δηλαδή για την εποπτεία της ε, μείωσης ε, των εκπομπών ρήπων, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι τα νέα θεσμικά όργανα τα οποία δημιουργήθηκαν με το Κανκούν να μπορέσουν να ε, αρχίσουν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, το Πράσινο Ταμείο για το Περιβάλλον το πλαίσιο του Κανκούν για τις προσαρμογές. Ε, η Επιτροπή επίσης προσαρμογής ε, και ε, τεχνικών, προδιαγραφών και του δικτύου. Εξακολουθούμε να ε, προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση για τη μεταφορά των ποσοστώσεων εκπομπών ρήπων, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο να μπορέσει να ολοκληρωθεί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας πρώτα απ' όλα και πρωταρχικά έγκυται στο ότι εμείς με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει να μπορέσουμε να διατυπώσουμε ποιες είναι οι επιμέρους θέσεις τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του Κανκούν. Ένα άλλο σημαντικό έργο θα είναι εμείς αποκινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, και στις ε, υψηλού επίπεδου διμερείς επαφές να εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πρέπει. Εκπροσώπηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και εκπροσώπηση των συμφερόντων επιπλέον και των κρατών μελών εξίσου. Η Ουγγρική Προεδρία θέλει να συνεχίσει προφανώς ε, το έργο της Βελγικής Προεδρίας ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα να προαχθούν αποτελεσματικά και δικός μας στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προπομπός, να είναι πραγματικά πρωτοπόρος στις διαπραγματεύσεις, διεθνείς διαπραγματεύσεις και να αναλάβει και ε, διαμεσολαβητικό ρόλο. Επίσης θα πρέπει οι διοργανωτές ε, της ε, νέας συνόδου για το κλίμα στην Νότια Αφρική να υποστηριχθούν ώστε στις προσπάθειές τους ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε μια, ένα πλαίσιο συμφωνίας στο Τέρμπαν. Πρέπει επίσης να συνεισφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να έχει ένα δικό της ξεχωριστό φιλόδοξο πρόγραμμα για τα κλιματολογικά θέματα και αυτό να μπορέσει να εφαρμοστεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολύ φιλόδοξη ακριβώς πολιτική για το κλίμα θα πρέπει να ακολουθήσει. Για να μπορέσει να προαχθεί αυτό το πρόγραμμα θα ήθελε η Ουγγρική Προεδρία να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει αυτό να γίνει πραγματικότητα. Ένα σημαντικός λοιπόν στόχος της, Ευρικής, της Ουγγρικής Προεδρίας, με συγχωρείτε, είναι οι διαπραγματεύσεις ε, για την πολιτική για τον άνθρακα σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ε, να μπορέσουν να προαθούν και να αριθμιστούν. Μετά το 2011 η στρατηγική για την μείωση του άνθρακα, της χρήσης άνθρακα θα προαχθεί. Θα πρέπει έτσι να οδηγηθούμε σε, μια, σε υψηλό ποσοστό ελεύθερη από άνθρακα οικονομία στην ανάπτυξή μας. Είναι ένα στρατηγικό έγγραφο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, προσανατολίζεται έντονα στην στρατηγική του 2020 όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Επίσης ε, συνδέεται και με άλλα στρατηγικά έγγραφα αυτό, για παράδειγμα με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, για παράδειγμα με το Energy Roadmap, τον οδικό χάρτη για τα ε, θέματα ενέργειας και τα συναφή ενεργειακά θέματα. Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης της χρήσης του άνθρακα και των ορυκτών καυσίμων πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθμίσουμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μερός τους στόχους μείωσης κατά 20% θα μπορούσε να, τους να αυξήσει αυτό το ποσοστό σε ένα υψηλότερο ποσοστό πάνω από το 20%. Να προωθήσουμε την ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη στρατηγική μεταξύ των κρατών μελών. Και μέχρι τέλη της Προεδρίας μας θα επιθυμούσαμε να είχαμε μια κοινή θέση του Συμβουλίου που θα καθιστούσε εφικτό να μπορέσουμε στη συνέχεια να περάσουμε με, από μια γέφυρα, από μια μεταβατική περίοδο προς μια νέα διαμόρφωση των οικονομικών θεμελίων της οικονομίας μας. Η στρατηγική απομάκρυνσης από τον άνθρακα και μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα έχει και ένα ορθολογικό πλαίσιο και στοχοθέτηση ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε όπως προαναφέρθηκε ένα στόχος πάνω από το 20% μείωσης. Αυτά τα θέματα πρέπει ε, σε άλλη σε συνάρτηση το ένα με το άλλο να εξεταστούν. Η Ουγγρική Προεδρία θέλει να διοργανώσει ομάδες εργασίας και συσκέψεις και ε, συνεδριάσεις που θα εξετάσουν και θα συζητήσουν τα διάφορα στοιχεία αυτής της στρατηγικής. Η πρώτη τέτοια ανταλλαγή απόψεων θα ακολουθούσε το Μάρτιο στη συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος. 24 έως 26 Μαρτίου θα έχουμε μια άτυπη υπουργική συνδιάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη όπου μια περαιτέρω προσέγγιση των διαφορετικών θέσεων θα ε, πρέπει να ε, γίνει ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της έκθεσης και το πώς θα συνεχιστούν αυτές οι ε, διαπραγματεύσεις θα μπορέσει πάλι να επαναγγραφεί στην ημερήσια διάταξη αυτό το ίδιο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Προεδρίας μας από πλευράς Ουγγλικής Προεδρίας του Συμβουλίου αυτό που θα θέλαμε είναι να προσπαθήσουμε τη συζήτηση να την θέσουμε στη σωστή τροχιά, στη σωστή πορεία. Κατά πόσον είναι ρεαλιστικός ο στόχος της μείωσης κατά 20% και θα δούμε και ποιους κινδύνους συνεπ πάγεται μια τέτοια πολιτική, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη διάσκεψη του Κανκούν είχε υιοθετήσει ένα ψήφισμα το οποίο έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι πρόθυμη και έτοιμη μονομερός ε, να προβεί χωρίς ε, κάποιες άλλες προϋποθέσεις και όρους σε ε, μια αύξηση του στόχου του 20% στο 30% της μείωσης ρήπων. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχει ακόμα συνένεση. Κάποια κράτη-μέλη υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα, κάποια άλλα όχι. Επίσης, το Συμβούλιο για το Περιβάλλον τον Οκτώβριο 2010 ζήτησε από το Συμβούλιο συνολικά να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις και μελέτες για το θέμα αυτό. Το Νοέμβριο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνταχθεί μια περαιτέρω μελέτη, μια περαιτέρω έκθεση για αυτό το θέμα και αυτό το θέμα να προετοιμαστεί υπό το φως των ε, ε, αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων του Κανκούν να επικαιροποιηθούν τα πράγματα και προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβληθεί μια περαιτέρω έκθεση τώρα κατά τη διάρκεια του έτους. Η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί πολύ σημαντική τη δυνατότητα μιας μείωσης πάνω από 20% όπως προανέφερα ήδη εκείνο το οποίο θα είναι η στρατηγική μείωση της χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2020 θα διαρκέσει ως χρονοορίζοντα και θα έχει και μεσοπρόθεσμους στόχους. Μπορούμε στη συνέχεια μετά ή να εκτιμήσουμε κατά πόσον θα ήταν δυνατόν μετά να ακολουθηθεί, να υιοθετηθεί ένα στόχος πάνω από το 20% που θα ενταχθεί στην πρόθεσμη στρατηγική σε έναν απότερο χρονορίζοντα και θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποια μέτρα είναι αναγκαία ώστε να έχουμε μια οικονομία η οποία θα βασίζεται σε μικρότερο βαθμό στον άνθρακα και τα ορικά καύσιμα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ένας φιλόδοξος στόχος μείωσης πρέπει να εξακολουθήσει να είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ω Ουγγρική Προεδρία να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Έτσι εξυπηρετούμε όχι μόνο τα δικά μας ουγγρικά συμφέροντα, αλλά συνεισφέρουμε στις παγκόσμιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών, που είναι τόσο σημαντική υπόθεση. Υποστηρίζουμε ακόμα και την πρωτοβουλία η, η πολιτική για το κλίμα και το περιβάλλον μέσα σε ένα πολιετές πλαίσιο προβλέψεων και προγραμματισμού να ενταχθεί. Είναι σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας τα αναγκαία κονδύλια, ώστε η πολιτική αυτή να προαχθεί όπως πρέπει. Εμείς ως Προεδρία του Συμβουλίου θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες ώστε πραγματικά να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το αναγκαίο χρηματοδοτικό οικονομικό πλαίσιο για την χρηματοδότηση αυτής της στρατηγικής μείωσης του άνθρακα των καυσίμων. Θέλουμε να συνεισφέρουμε ενεργά όσο περνάει το χέρι μας. Τέλος, καταδεικνύεται ότι η Ουγγρική Προεδρία έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την Προεδρία της που προσανατολίζεται ιδιαίτερα έντονα στου προσανατολισμού για την προστασία του περιβάλλοντο και τη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Συνεχίζεται η πορεία τη Βελγική Προεδρία και συνδέεται το έργο μα με την επόμενη Προεδρία που θα είναι τη Πολωνία, ώστε από κοινού να εξυπηρετήσουμε του κοινού μα στόχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και εσείς κύριοι Ευρωβουλευτές να μας υποστηρίξετε. Χωρίς μια ενεργό τέτοια συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων η Ουγγρική Προεδρία δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εκθέσαμε. Και γι' αυτό θα θέλαμε ε, συνεχώς να συνεργαζόμαστε μαζί σας και να διαβουλευόμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ για την προσοχή. vielen Dank, Herr ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την παρουσίαση του προγράμματός σας. Νομίζω ότι το Υπουργείο σας έχει μια πολύ καλή δομή και για την ανάπτυξη των περιοχών, περιφερειών, των δήμων, κοινοτήτων σε συντονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος είναι μια σύγχρονη ε, ας το πω δομή οργανωτικά που έχει δυνατότητες να αποδώσει στο μέλλον. Ακούσαμε προσεκτικά για τους επόμενους μήνες αυτά που μας είπατε για τη στρατηγική σας για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής και στη Νότια Αφρική αλλά και για μια αυτόνομη πολιτική και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς μας. Γνωρίζουμε όλοι το 2005 ποιο είναι ποιοι είναι οι στόχοι μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα έχει αποφασίσει αυτά τα πράγματα ήδη. Τώρα θέλουμε τα ενδιάμεσα βήματα να καθοριστούν και να προσδιοριστούν. Να μην χάσουμε χρόνο, να μην χάνουμε περαιτέρω χρόνο. Και όταν φυσικά αυτή τη δεκαετία πρέπει να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε γιατί διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας του 2050 αν δεν το κάνουμε αυτό. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται με τις πολλές ερωτήσεις που έχουν ζητηθούν να διατυπωθούν, έχει ζητηθεί να διατυπωθούν. Μέχρι παρατέτατο θα έχουμε χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι 1,5 λεπτό καθένας ε, για ερωτήσεις σχόλια. Ξεκινάμε με τον Ρίχαρτ Ζέμπερ για το ΕΛΚ. Παρακαλώ κύριε Ζέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι Υπουργέ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Θέλω να ε, συγχαρώ και ο ε, Πέτρο Λάιος είχε έρθει ως υφυπουργός στη δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή ε, που έδωσε σημαντικές μάχες για το κλίμα. Θέλω κάποιες ερωτήσεις να θέσω. Παρουσιάσατε ένα ωραίο πρόγραμμα. Εκείνο το οποίο απουσιάζει κάπω για μένα είναι μπορείτε να είσαστε πιο εξειδικευμένο όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Διότι αυτά τα μέτρα όλα θα συνδέονται με κόστη και δαπάνε. Και για κάποια κράτη-μέλη, χωρί να κατονομάσω κάποια, ίσω και για κάποια τα οποία έχουν ε, ε, κορβανά, πλήρη, γεμάτο και συνεισφέρουν ως χορηγοί, ενδιαφέρει άμεσα αυτό. Ποιε θα είναι οι δαπάνε για τα προβλήματα του σημερινού συστήματος. Πουλάνε αερακοπανιστό πολλά από τα κράτη σήμερα. Υπάρχουν τα προβλήματα και χρειάζονται πραγματικά μέτρα για την προστασία του κλίματος. Πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Δεύτερον, για τη χρηματοδότηση. Αναφέρατε το Κανκούν. 100 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 αποφασίστηκε να δαπανηθούν. Τεράστιος όγκο χρημάτων αυτός και για την ιδιωτική οικονομία. Ποιες προτάσεις έχετε για να καλυφθούν τα κόστη. Μια και είσαστε υπουργό Φυσικών Πόρων και βλέπουμε ότι αυτά και σε σχέση με, τη, ε, με το νερό, με τους υδάτινους πόρους, τι θα γίνει. Είσαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει. Τι θα προτείνατε. Ευχαριστώ. Ο Ρίχατς Πάπας για τα θέματα των υδάτινων πόρων αλλά και για τον Σάντορ Φαζάκα, ε, στο επόμενο Υπουργό θα μπορούσε να τεθεί αυτό το ερώτημα για τους υδάτινους πόρους θα μπορούσαμε για το δεύτερο γύρο να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Συνεχίζουμε. Ματία Ρότε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για το γεγονό ότι είσαστε εδώ, για το ότι μα παρουσιάσατε το πρόγραμμά σα για τι διεθνεί διαπραγματεύσει του Κανκούν, που ήταν καλύτερε από ό,τι αναμέναμε, αλλά χειρότερε από ό,τι ελπίζαμε. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα πακέτο για το κλίμα και έχουμε διαφορετικού τομεί. Ε, και για τον τομέα των ενέργειων μεταφορών όμω ε, εξακολουθεί να υφίσταται ότι μια ε, διεθνής οργάνωση εκεί ε, τροχοπέδησε τα πράγματα και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και ο ναυτιλιακός ε, τομέας να συμπεριληφθεί στις εκπομπές ρήπων και να συνυπολογίζεται η Διεθνής Οργάνωση, ο Οργανισμός ο Διεθνής του ε, ΟΗΕ και η IMO εμπλέκεται και έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναμένει μια προθεσμία μέχρι τα τέλη του 2011 για να υποβληθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερώτησή μου, ποιες τομεακές προτάσεις μπορούμε να αναμένουμε υπό την Ουγγρική Προεδρία και για τον στόχο ε, του, του 30% στην ανάλυση του συμπεριλάβαμε εμεί ένα μεγάλο πακέτο για το κλίμα και αν συμμετάσχουν τα άλλα μεγάλα κράτη θα μπορέσουμε να έχουμε μείωση 30%. Μπορείτε να μας επεξηγήσετε τι γίνεται με τη μείωση αυτή και με την, ε, ε, τις μεταβολές που θα συνεπάγεται και αυτό στην ανάλυση σας να ενταχθεί. Κατά το πρώτο εξάμεινο αυτού του έτους θέσαμε ενώπιον μας το στόχο να καταφέρουμε να έχουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που θα συντάξουμε. Θα με ενδιέφερε λοιπόν να μάθω πώς αυτός ο στόχος συγκεκριμένα συζητείται στο Συμβούλιο, γιατί μέχρι σήμερα ήταν, μέχρι τώρα ήταν κάπως γενικόλογες οι αναφορές αυτό. Ευχαριστώ. Ρίτα Μάνας παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ουγγρό Υπουργό επίσης. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας παρουσίαση του προγραμματός σας. Η ερώτησή μου σχετίζεται με τα οικοδομικά υλικά, ε, διότι όταν ομιλούμε ε, για τον περιορισμό ε, των εκπομπών άνθρακα ή της χρήσης άνθρακα, το ξύλο παραδείγματος χάρη είναι ένα ανανεώσιμος πόρος και μπορεί να, επανα, να ανακυκλωθεί. Τα δέντρα φυτρώνουν και μεγαλώνουν στα δάση. Τα δάση θα πρέπει να διατηρηθούν και ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των δασών ώστε να διαχειριστούν σωστά τα δάση. Να τα, η, η, σήμανση όσον αφορά το περιβάλλον είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια, ένα εναρμονισμένο σύστημα σήμανσης. Και το δεύτερο ερώτημά μου αφορά τους στόχους ενεργειακής ε, απόδοσης. Ε, το ξύλο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις, ε, στις κατασκευές. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ενεργειακή απόδοση αλλά και τον κύκλο ζωής των υλικών που χρησιμοποιούνται για, την, για τις κατασκευές. Ευχαριστώ. να δει ότι οι συνάδελφοι προέρχονται από ένα ε, μια χώρα που έχει μεγάλα δάση. Η ερώτηση αυτή θα πρέπει να διαβιβαστεί και στο συνάδελφο Φασέκας που θα έρθει υστερότερα, που είναι αρμόδιος για θέματα δασοκομείας, δασοπονίας. Αυτός θα μπορούσε να απαντήσει την ερώτηση. Και τώρα η επόμενη παρέμβαση, εσείς παρακαλώ. Uh, θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Υπουργό στο Κοινοβούλιο. Οι πράσινοι προσπαθούν να έχουμε ένα πρόγραμμα εργασίας ιδιαίτερα φιλόδοξο για τα θέματα του περιβάλλοντος. Το βασικό πρόβλημα τους επόμενους μήνες είναι να κλείσουμε την διαφορά ανάμεσα στους δύο, στο στόχο που έχουμε για τους δύο βαθμούς μείωση και τις διεθνείς ανηλυμένες μας υποχρεώσεις. Το θέμα είναι πώς θα κλείσουμε την απόσταση ανάμεσα στα δύο. Βλέπουμε ότι ε, είχαν ξεκινήσει θα έχουν ξεκινήσει μάλλον κάποιες ενδιάμεσες εκλογικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ξεκινήσει η συνάντηση του Ντέμπαν, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με τις αναδυόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, της Ινδίας, ε, της Κίνας κτλ τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεργαστούμε και να πείσουμε τις χώρες αυτές. Τώρα για τις δικές μας ανηλυμένες υποχρεώσεις, όταν ζητάμε από άλλες χώρες να κάνουν κάποια προσπάθεια, πρέπει και εμείς να κάνουμε μια αντίστοιχη προσπάθεια. Με χαρά άκουσα ότι εσείς στο Συμβούλιο του Ιουνίου θα βγάλετε κάποια συμπεράσματα που θα οδηγούν στο 30%. Υπάρχει επίσης το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας της ενεργειακής. Έχουμε μείνει πίσω πρέπει να έχουμε κάποιους δεσμευτικούς στόχους προ την κατεύθυνση αυτή. Πώς μπορεί η Ευρώπη να κρατήσει τι υποχρεώσει, να σεβαστεί τι υποχρεώσεις της και πώς αυτό θα φαίνεται στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. για, για την Ενωτική Αριστερά παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω θερμά και στον Υφυπουργό σα και πρώην συνάδελφό μα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη διεθνή ατζέντα επίση. Είπατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση και υπογραμμίσατε την ανάγκη της νομικής δέσμευσης και ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους περιλαμβανομένων και των αναδυόμενων οικονομιών. Αυτό που λείπει από τη γλώσσα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, που πρέπει και αυτοί να εφαρμόσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Πώς λοιπόν ε, θα γίνει αυτή η συνεργασία με τις αναδυόμενες οικονομίες ε, και τις Ηνωμένε Πολιτείε εν ώψη του Ντέρμπον και ποια είναι η ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά την Ινδία και πώς θα βοηθήσουμε τη θέση του κυρίου Ράμος ο οποίος προσπαθεί να παίξει έναν θετικό ρόλο και γνωρίζουμε τις δυσκολίες που δημιουργούνται στην χώρα του. Ε, ακριβώς λοιπόν πώς οι αναδυόμενες οικονομίες θα ε, τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Θα ήθελα επίσης να συνδέσω το ερώτημα ε, με το 20% και την ανάγκη να είναι και αυτός ένας δεσμευτικός στόχος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν είναι πολλοί συνάδελφοι εδώ παρόντες. Παρόλα αυτά όμως Υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει από πλευρά των συναδέλφων. Δεν ξέρω αν έχει αρκετό χρόνο ο υπουργό μέσα σε 20 λεπτά να απαντήσει τόσε πολλέ ερωτήσει. Και εγώ θα είχα μια ερώτηση για το θέμα του πρωτοκόλου του Κιώτο. Για το μέλλον του πρωτοκόλου του Κιώτο έκανε λόγο ο ίδιο ο Υπουργό πιο πριν. Συχνά το έχω αναφέρει εδώ στη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική μα Επιτροπή και έχω πει ότι είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα υφίσταται μεταξύ των νέων και των παλαιότερων κρατών μελών και ένα πρόβλημα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιπλέον και πολλών Ευρωβουλευτών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι υπόψη της. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι οι <clears throat> ποσοστώσεις για το διοξίδιο του άνθρακα <clears throat> μετά το 2012 να μην δημοπρατούνται, να μην πολλούνται. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό για τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχική, Δημοκρατία της Τσεχίας και άλλες ε, χώρες που πλήρωσαν αντίτιμο για να υπογραφεί το, ε, η Συμφωνία του Κιώτο. Υλοποιήσαμε και υπερυλοποιήσαμε, ε, υπερ, καταφέραμε σε πλήρη και υπερπλήρη βαθμό να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Και τώρα τι θα γίνει. Χωρίς εμάς δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει τους στόχους. Η Ουγγρική Προεδρία πρέπει αυτή την τροχοπέδηση τώρα να την άρει. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να προχωρήσουμε. Θα είναι σε θέση η Ουγγρική Προεδρία να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, ώστε οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες, μια και υποχρεώθηκαν, αν μετά το 2012 θα δημοπρατούνται αυτές οι ποσοστώσεις, θα μπορούν να αγοράζονται ποσοστώσεις, μόνο υπό συγκεκριμένους όρους να μπορούν να γίνουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσία του. Θα ήθελα να επιστρέψω λίγο, λίγο πιο πίσω μάλιστα. Δεν έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το κλίμα εάν δεν δώσουμε μια σαφή απάντηση στην λεγόμενη κοινή αλλά διαφοροποιούμενη ευθύνη, την δήλωση του Μπαλί δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Θα πρέπει επίσης να δούμε την δυνατότητα αποδοχής κάποιων ορίων τα οποία να είναι νομικά δεσμευτικά. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται σε σύγκρουση αν θέλετε με την έννοια της απόλυτης κυριαρχίας. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς ζούμε κάτω από ορισμένες συνθήκες τις οποίες θα χαρακτήριζα συνθήκες αλληλοεξάρτησης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές αλλαγές. Προ την κατεύθυνση αυτή λοιπόν θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχουν πολιτικές προτάσεις για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το ε, αδιέξοδο. Ένα δεύτερο θέμα αφορά την προσαρμογή στις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών. Εμείς προσπαθούμε στην Steering Committee, στη Διευθυντική Επιτροπή για την Κλιματολογική Αλλαγή, να υιοθετήσουμε μια πρόταση πολιτική επεξεργασίας των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Λίζε, ο οποίος θέλησε να μάθει αν ταιριάζει σε αυτό το χαρτοφυλάκιο η αποδοτικότητα της χρήσης ενεργειακών πόρων. Ναι, ταιριάζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να συμβεί και με εμένα, όπως και με άλλους συναδέλφους, να διαβιβαστεί, λέει, υστερότερα σε άλλον η ερώτησή μου. Ήμουν εγώ συντάκτη ε, έκθεση για το θέμα τη ε, αποδοτική εκμετάλλευση ενέργεια και στην επόμενη σύνοδο ε, θα ενταχθεί αυτό το θέμα και ανησυχώ για αυτά τα οποία θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε υπέρ δεσμευτικών στόχων. Ρεαλιστικό δεν θα είναι τόσο αυτό να, ότι θα υπάρξει λύση όπως το φαντάζεται και το επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Εντάξει, όμως ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες έχω επειδή προδιαγράφεται και μετά από διαφορετικές συζητήσεις το βλέπουμε αυτό ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν θα επομισθούν ευθύνε για αυτό το στόχο και θα δώσουν την εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη να αναλάβει τη ρύθμιση. Τώρα, ένα σε σχέση με, το, με αυτό το θέμα, ε, και την, έχουμε την δέσμευση έναντι των ε, ψηφοφόρων μας ε, και το 70% σε σχέση με τη Γερμανία για παράδειγμα. Το θέμα είναι στα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε όχι μόνο ρύθμιση αλλά και κίνητρα να δημιουργήσουμε φορολογικά κίνητρα, πιστώσει, δάνεια, ώστε να να κινητοποιηθούν οι πολίτες με αυτά τα κίνητρα να κινηθούν προς την αποδοτικότητα της ε, ενέργειας, τότε κάτι πρέπει να γίνει από εσά. Ζητώ πριν από το Συμβούλιο, πριν από τη Σύνοδο να αναφερθεί ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δηλώσουν δεσμευτικά ότι θα κάνουν και εκείνα κάτι και δεν θα περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν ρυθμίσεις. Δηλαδή δεν θα είναι δημοφιλέ να έχουμε μόνο ρυθμίσεις και να μην κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σνερχάτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Ουσιαστικά για μένα πρόκειται για τα μέσα χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή τη συζήτηση επανειλημμένα την είχαμε, ότι εδώ αναφερόταν και λέγατε ότι εδώ προκαλούμε ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες δημιουργείται φτώχεια και προξενούμε αυτή τη φτώχεια. Τα συζητάμε και στη συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ συνολικά και σφαιρικά. Κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε όμως και θα ήθελα να μάθω τι σκοπεύει να κάνει η Ουγγρική Προεδρία ώστε αυτή η δυνατότητα υποστήριξης αυτών των χωρών για τις κλιματικές αλλαγές ποια νέα μέσα θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το στόχο και δεύτερο έχουμε ήδη, έχουμε ήδη στην διαπραγμάτευση ε, για την εμπορία ε, διαπραγμάτευση εμπορίας τρύπων κάποια προβλήματα. Υπάρχουν και εγκληματικές πράξεις που έχουν σημειωθεί κάποια πιστοποιητικά συντάσσονται και πολλούνται ενώ τίποτα δεν κρύβεται πίσω από αυτά, ε, δεν υπάρχουν ερίσματα και Χρήματα διακινούνται έτσι. Ερώτηση, πώς θα επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται ένα νέο σύστημα ή πρέπει να επανορθωθεί το παλαιό. Ευχαριστώ. Καλή ερώτηση λέει ο Πρόεδρος. Και μια καλή απάντηση θα δοθεί σίγουρα σε αυτήν την καλή ερώτηση. γιατί τη χρηματοδότηση αναφέρατε εσείς πιο πριν ότι η προστασία του κλίματος και στην μεσοπρόθεσμη, στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για τα οικονομικά, για τα κονδύλια θα πρέπει να διαδραματίζει ένα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω αυτό το θέμα. Ερώτηση, έχετε υπόψη ένα ξεχωριστό κονδύλιο στον προϋπολογισμό που θα εμφανίζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, διότι πολλά κράτη-μέλη αγωνίζονται για την χρηματοδότηση της προστασίας του, κλίματο. Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για την προστασία του κλίματο θα μπορούσε να είναι πολύ επικοδομητικό. Ξέρουμε να υπάρξει κάποιο κίνητρο, κάποια πρόθεση ώστε να μπορέσει αυτό να διασφαλιστεί και έτσι θα είναι στην pipeline καθοδόν ε, υπό εξέλιξη αυτό ώστε στην, ε, στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη. Πολλές ερωτήσεις είχατε, 10 λεπτά ίσως ε, και ίσως μπορείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να απαντήσετε παρακαλώ. Πολύ σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω εκ προημίου κάτι. Θα ήθελα να πω ότι είναι προφανές ότι εγώ επί της ουσίας αυτές τις ερωτήσεις όλες μέσα σε 10 λεπτά δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες. Ελπίζω ότι τους επόμενους 6 μήνες θα έχω την δυνατότητα να διαβουλευτώ μαζί σας, να συνεχίσω την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για να μπορέσουμε να τα δούμε καλύτερα αυτά. Είμαι και πρόθυμος να συμμετάσχω και σε μια ακρόαση αν το επιθυμείτε. Θα θέλαμε επίσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας μέσα στο πλαίσιο μιας ε, υποβολής έκθεσης προόδου να σας εκθέσουμε τα σχετικά. Ποιους στόχους δηλαδή μεταξύ καταφέραμε να πετύχουμε από αυτούς που εντάσσονται στο πρόγραμμά μας. Πιστεύω ότι αμφότεροι το χρειαζόμαστε αυτό. Μία έκθεση πρόοδου. Μία έκθεση ποια πρόοδο σημειώνεται. Θα ήθελα εκ προημίου να ζητήσω συγγνώμη, διότι μόνο πολύ σύντομα κάποιε ερωτήσει θα μπορούσα να απαντήσω και όχι σε βάθο. Όσον αφορά την χρηματοδότηση. Εδώ όμω να προσθέσω και κάτι. Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε και γραπτές, γραπτός απαντήσεις. Όσον αφορά την χρηματοδότηση όπως έλεγα. Εδώ υπάρχουν αρκετές πολλές πτυχές. Στο Κανκούν ελήφθη μία απόφαση για την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και ένα, την άμεση έκθεση για την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τα συναφή. Εμείς θα πρέπει το πράσινο ταμείο για το περιβάλλον να καταφέρουμε μετά τον Τέρμπα να, αφού θα έχει δρομολογηθεί να λειτουργήσει και σωστά. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ορθή αποτελεσματική επικοινωνία. Όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση θέλουμε να οικοδομήσουμε στην προσπάθεια δημιουργία ενό κλίματο εμπιστοσύνη. Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο πλαίσιο χρηματοδότηση, ήδη στην Κοπενχάγη υπήρξε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία οι, αναπτυσσο... οι αναπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020 θα έπρεπε να δημιουργήσουν ένα ταμείο με περίπου 100 δις δολάρια στο Κανκούν τα συμβαλόμενα μέρη συμφώνησαν αυτά τα 100 δις δολάρια από τους πιο διαφορετικούς τομείς να συναπαρτίζονται, να συντίθενται. Θα υπάρχουν κονδύλια και αυτό ο ίδιος ο πρόεδρος το ανέφερε, ο πρόεδρος ε, στον Ουγγρικό για παράδειγμα προϋπολογισμό έχουμε ξεχωριστό ε, κεφάλαιο, ξεχωριστή κατηγορία κονδυλίων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ήδη μια πρόοδος. Και επιπλέον εδώ και διμερός αλλά και πολυμερός ε, θα υπάρξουν κονδύλια που θα διασφαλιστούν και εναλλακτικά κονδύλια. Πέρα από αυτό είναι σημαντικό θεωρούμε κονδύλια από την ελεύθερη αγορά να μπορέσουν να συλλεγούν και να συσσωρευτούν. Πρόκειται για μακροπρόθεσμους στόχους και χρονοορίζοντες. Πρόκειται για διαθωτικές μεταβολές που θέλουμε να επιτύχουμε. Η Διαρκής Επιτροπή, η Μόνιμη Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση των Κλιματεολογικών Κλιματικών Μέτρων πρέπει να διασφαλίσει ότι θα βελτιωθεί ο συντονισμός και η χρηματοδότηση Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές ροές και διεργασίες θα είναι πιο αποτελεσματικές και να κινητοποιηθούν και οι πόροι. Επιπλέον το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική υπόθεση να καταφέρουμε μια και την ερώτηση αυτή την διατύπωσαν αρκετοί ευρωβουλευτές, να δούμε ότι η κλιματική πολιτική συνδέεται με τα θέματα ενέργειας και τα θέματα μεταφορών και αυτά κατά τη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας θα πρέπει να αντανακλώνται στη δράση μας. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στον προϋπολογισμό και σημαντικές επιπτώσεις ε, στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό μετά το 2013. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για θεμελιώδη στρατηγικά ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητα, συγκεκριμένοι τομείς ε, στο κλιματικό τομέα και στην ενεργειακή πτυχή να ληφθούν υπόψη στη χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών να μπορούν να καλύπτονται αυτές οι συνιστώσεις. Στη χρηματοδότηση των επενδύσεων για παράδειγμα μέσα σε όλο αυτό το σφαιρικό πλαίσιο δημιουργούνται ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν. Αυτά είναι τα πιο κέρια, τα πιο κρίσιμα σημεία. Πρόκειται για την ενεργειακή μας πολιτική, για την πολιτική μας για τις μεταφορές, για την χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών μας. Πρόκειται επίσης για το ότι συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στο πλαίσιο του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και του Πράσινου Ταμείου. Είναι διαφορετικά θέματα που μας απασχολούν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και θα διαδραματίσουν και σημαντικό ρόλο και στις ε, ιστερότερες συζητήσεις. Όλα αυτά αλληλοσυνδέονται οι διάφοροι, τομείς και τα τομεακά θέματα πρέπει σε ένα ενιαίο πλαίσιο σφαιρικά να αντιμετωπιστούν. Οι νέε δημοσιονομικές προοπτικές τώρα προετοιμάζονται και σχεδιάζονται και θα πρέπει οπωσδήποτε στην προκατακτική αυτή φάση να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. αφορά το νερό, του υδάτινους πόρου, την πολιτική μας για τους υδάτινους πόρους. Εν μέρη θα ήθελα εγώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Μερικά όμως εν μέρη είναι αρμοδιότητα του ε, Υπουργού μας ε, Φεζεκάς και αυτός πιο εξειδικευμένα θα μπορέσει στη συνέχεια υστερότερα να σας απαντήσει. Εδώ θα ήθελα εγώ να αναφέρω ότι η στρατηγική για τον ποταμό Δούναβη έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Είναι αυτό ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για του υδάτινους πόρου. Η πολιτική για τον Δούναβη είναι μόνιμο στοιχείο της Ουγγρικής Προεδρίας. Η Ουγγαρία ασχολείται φυσικά με τη συνάφεια και τη συνάρτηση μεταξύ κλιματικών αλλαγών και υδάτινων πόρων. Οι Ούγγροι ειδικοί και πραγματογνώμονες επιβεβαιώνουν τις επιφυλάξεις που υφίστανται και όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και που τις έθεσαν αυτές τις επιφυλάξεις στο Κανκούν. Είπαν οι αναπτυσσόμενες χώρες ότι η υδάτινη πολιτική για τα ύδατα πρέπει να ενταχθεί μέσα στη σφαιρική πολιτική για την προστασία του κλίματος. Πρέπει εδώ να πετύχουμε σωστή ισορροπία για τους υδάτινους πόρους και για τον κύκλο, ας το πούμε έτσι, των ε, ε, κλιματικών ζητημάτων και της μετανάστευσης που θα προκληθεί αν υπάρξουν προβλήματα. Η έκθεση για τις κλιματικές αλλαγές κάνει λόγο για το πόσο σημαντική είναι η πολιτική για τους υδάτινους πόρους. Αν στη σημερινή, στη ήδη κατάσταση μπορεί, να υπάρξει ε, λειψιδρία και μπορούν οι εισοδιές από τη Γεωργία να συρρυκνωθούν. Για παράδειγμα στην Αφρική, στην ε, ε, Νοτιοανατολική Ασία, στην ε, Νέα Ζηλανδία. Και αυτά όλα θα δημιουργήσουν, δημιουργούν προβλήματα στην κεντροανατολική Ευρώπη πολλές φορές ε, κατά τη διάρκεια του θέρους υπάρχει λειψιδρία, υπάρχει ανομβρία λειψιδρία. Η ξηρασία αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε την ευαισθησία των κρατών, την, ε, με ε, τον ευάλωτο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον ε, ε, περιορίσουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα διαπεριφερειακά και περιφερειακά για την πολιτική για τους υδάτινους πόρους που θα στοχεύουν στο να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Γκρότε αναφέρθηκε στις εναέριες μεταφορές και στις ε, ναυτιλιακές μεταφορές και αναφέρθηκε στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από αυτούς τους τομείς και τη συμπερίληψή τους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αναμένει την υποβολή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ουγγρική Προεδρία και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωβουλή, μαζί σας δηλαδή, θα υποβάλουμε εμείς ως Ουγγρική Προεδρία προτάσεις για αυτά τα θέματα στο ε, σώμα εκπροσώπων των ε, πραγματογνωμόνων. Όσον αφορά το carbon leakage, την ε, διαρροή άνθρακα, διαφυγή άνθρακα, αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Ιδιαίτερα για τις μεθοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ουγγαρία ειδικότερα. Βλέπουμε ήδη ίχνη και αποτυπώμα, ε, σημάδια αυτού του προβλήματος και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχει μετακίνηση από την Ουγγαρία για παράδειγμα προς την ε, Ουκρανία. Αυτά μπορούν να δημιουργούν προβλήματα, δημιουργήσουν προβλήματα μεθοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τα υλικά, για τις οικοδομές. Ε, τι θέθηκε ένα θέμα για αυτό το ζήτημα από έναν Ευρωβουλευτή. Έχουμε και θέματα εδώ δασοκομείας ε, και δασοπονίας. Ο συνάδελφός μου Φέζεκας, Ούγγρος Υπουργός στη συνέχεια απαντήσει αυτό, αυτά τα, αυτές τις εξειδικευμένες πτυχές. Για την υλοτομία και την δασοκομεία είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Πρέπει να μιλήσουμε, να κάνουμε λόγο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπό αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικά τα δάση. Βασιζόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπολογίζουμε σε αυτές για τα προγράμματα αποδοτικότητας, ενεργειακής αποδοτικότητας. Ένα παρόμοιο, ένα συναφές τέτοιο ε, ζήτημα αφορά τις, ε, κλιματικές, τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα με τις ΗΠΑ και τις αναδυόμενες χώρες, ε, τρίτες χώρες δηλαδή. Βραζιλία, Ινδία, Κίνα κτλ. Ετέθη ένα ερώτημα ήδη για αυτό το θέμα. Πώ αξιολογούμε εμεί αυτό το ζήτημα, ποιε είναι οι σχέσει μα με αυτέ τι χώρε και ποια επιχειρήματα χρησιμοποιούμε εναντί αυτών. Προσέξτε, οι διαπραγματεύσει για αυτό το θέμα διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο των, ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Εθνών εξαρτάται από το πώ αυτές οι διαπραγματεύσει στα Ηνωμένα Έθνη θα προαχθούν, από ποια πρόοδο θα σημειώσουν για να πούμε ποια, τι θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συνεργαζόμαστε ω Προεδρία με την κυρία Χέντεγκαρντ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχουμε στην προπαρασκευή αυτών των συνεδριάσεων και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το οποίο ήδη προανέφερα στην εισαγωγή μου, ποιες προτεραιότητες έχει η Ουγγρική Προεδρία σε σχέση με τα κλιματολογικά θέματα. Αυτές τις προτεραιότητες επιθυμούμε εμείς να υλοποιήσουμε και να επιτευχθούν. Θέλουμε να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν οι προτεραιότητες αυτές, οι στόχοι που θέσαμε και να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Προσπαθούμε λοιπόν τις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως τους μεγάλους εκπομπούς ρήπων, ε, τις χώρες που έχουν υψηλές εκπομπές ρήπων, να μπορέσουν αυτές οι αρχές να, υιοθετηθούν και από αυτές τις ανα, αναδιόμενες, αναψώμενες χώρες. Αν δεν το καταφέρουμε να υιοθετηθούν αυτοί οι στόχοι από αυτές τις χώρες, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ένα στόχος σημαντικός είναι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε δύο βαθμούς Κελσίου. Προαναφέρθηκε αυτό από συνάδελφό σα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα υποβληθεί μια πέμπτη έκθεση για τις κλιματικές αλλαγές του του IPCC και μέσα στο πλαίσιο αυτής της πέμπτης έκθεσης θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε επικίνδυνες τέτοιες κλιματικές αλλαγές και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις μπορούμε να προλάβουμε και να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη. Οι αποφάσεις του Κανκούν εκινούν από το ότι η αναθεώρηση και επανεξέταση των συνολικών στόχων θα πρέπει να ξεκινήσει το 2013. Με αυτή την επανεξέταση πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διεργασίες μέχρι το 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την επανεξέταση, αναθεώρηση θα διαδραματίσει ένα σημαντικό σημαντικό ρόλο. Θέλουμε να καταστήσουμε, ε, να συνειδητοποιήσουμε, να γίνει ε, από όλου ε, να υπάρξει ευαισθητοποίηση ότι αν δεν τα καταφέρουμε θα μείνουμε πολύ πίσω από τις εξελίξεις και δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Επιπλέον, κάτι το οποίο σε πολλές ερωτήσεις βρήκε απήχηση και αναφέρθηκε, είναι ότι εμείς στις διαπραγματεύσεις για τα θέματα τα ενεργειακά και της ενεργειακής πολιτικής υφίστανται πολλές και μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη δεν συμφωνούν να υπάρχουν νομικά δεσμευτικοί στόχοι που θα υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τις επιδόσεις και τους στόχους. Η δική μου λοιπόν εντύπωση πρέπει να σας πω είναι, εγώ συμμετείχα βέβαια σε αρκετές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις προπα... προετοιμάζοντας την Ουγγρική μας Προεδρία. Η δική μου εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών τον, τους νομικά δεσμευτικούς στόχους ε, και τα πλαίσια αυτά μέσα στο πλαίσιο της ε, αποδοτικότητας ενέργειας δεν υποστηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν και νομικά δεσμευτικοί στόχοι όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Δεν την υποστηρίζουν λοιπόν. Θα είναι φυσικά όμως σημαντικό αυτή η στόχη νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα να δούμε ότι θα μπορούν να είναι χρήσιμοι εποφελής. Είναι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτούς τους νομικά δεσμευτικούς στόχους και μετρήσιμους στόχους ότι τους υποστηρίζει έναν των κρατών μελών που δεν τους υποστηρίζουν. Παρ' όλα αυτά είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών για διαφορετικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους αλλά και άλλους λόγους δεν υποστηρίζει η πλειοψηφία των κρατών μελών αυτή την πορεία κατά την διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, κατά την διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, μπορούμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να μεταπιστούν τα κράτη-μέλη. Έχω όμως αμφιβολίες αν μπορούμε να σημειώσουμε κάποια σημαντική μεταβολή, κάποια σημαντική αλλαγή μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες. Πολύ σύντομα τώρα, μια και έχω ίσως ένα λεπτό αν επιτρέπετε ακόμα, να πω δύο λόγια για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κύριος Σνέρχαντ έθεσε αυτό το ερώτημα. Πρόκειται για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πρόκειται για την χρήση νέων μέσων και εργαλείων. Μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και μέσων, νέων μέσων μπορούμε να υποστηρίξουμε την εξέλιξη, την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Μόνο εν μέρη πρόκειται για οικονομικά θέματα και μόνο εν μέρη προωθούμε και μπορούμε να στηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες με χρήματα. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί υποστήριξης και συνδρομής που δεν συνδέονται με κονδύλια ή με θέματα οικονομικά. Σε αυτές τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές και με, ε, προσαρμογές. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται εν μέρη επενδύσεις και χρήματα, κονδύλια αυτές οι χώρες, αλλά εν μέρη όχι. Όσον αφορά το, το πρωτόκολλο του Κιώτο, συμφωνώ με τον συνάδελφό σας. Πρέπει να βρούμε μια λύση για τα θεμητά νομιμοποιημένα αιτήματα και διεκδικήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι αυτονόητο ότι βέβαια υπό το φως της επίτευξης των στόχων μας πρέπει να γίνει αυτό. Μπορεί να είναι μείζον πρόβλημα για αυτές τις χώρες όταν το πρωτόκολλο του Κιώτο δεν την χάνει νομικά δεσμευτική συνέχεια. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό πρόβλημα. Γι' αυτό ασχολείται σε βάθος η Ουγγρική Προεδρία διεξοδικά με αυτό το ζήτημα. θα μπορούσα τώρα να σας αναφέρω ότι φαίνεται ότι δεν απάντησα μία ερώτηση. Ο κύριος Πρόντι μου έθεσε μία ερώτηση και δεν την απάντησα από ό,τι φαίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Πρόκειται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, η Ουγγρική πολιτική, η Ουγγρική Προεδρία καλύτερα, έχει μια παρόμοια προσέγγιση όπως εκείνη στο θέμα των ε, κονδυλίων των δημοσιονομικών Συμφωνούμε λοιπόν εμείς οι Ούγγροι στην Ουγγαρία με το ποσοστό των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το αυξήσαμε και μέσα στο ενεργειακό συνολικό μείγμα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία αύξησης του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει νέες δυνατότητες να υποστηρίξουμε. Για παράδειγμα το υδρογόνο αυτές τις νέες λύσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας διασφαλίσω κύριοι Ευρωβουλευτές ότι η ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα είναι για μας να συνεργαστούμε και να συνεχίσουμε συνεργασία όταν θα έχουμε χρόνο θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ Πρόεδρος, ευχαριστώ, ευχαριστώ εσάς κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Θα έλεγα εσείς και ο Υφυπουργό κ. Πέτερ Ολάγιο θα είσαστε πάντα στη διάθεσή μα όταν θα συνεχίσει αυτέ τι συζητήσει στο Κοινοβούλιο. Ο εισηγητή μα για την έκθεση 20% μείωση ε, του ποσοστού ε, διοξιδίου του άνθρακα ή και παραπάνω ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένο ότι θα υπάρξει συμμετοχή από πλευρά σα στι ακροάσει μα. Ε, θα έχουμε μια τέτοια ακρόαση. Αν επιθυμείτε, είσαστε ήδη προσκεκλημένος στην πρώτη μα ακρόαση για αυτό το στρατηγική σημασία θέμα. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Είμαστε ικανοποιημένοι να συνεχίσουμε συνεργασία μαζί σας και προσβλέπουμε στην Ουγγρική Προεδρία στους επόμενους έξι μήνες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, επιστρέφουμε στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε το σημείο 30. Έχουμε 30 σημεία στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε μία επιπλέον λοιπόν ανταλλαγή απόψεων με την Ουγγρική Προεδρία θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης Υπέθρου της Ουγγαρίας, τον κύριο Ζαντόρ Φαζέκας, που ασχολείται με θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και με την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι δύο από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Έχουμε ήδη συζητήσει θέματα που αφορούν την ε, δασοκομική δραστηριότητα, τη διαχείριση των δασών τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επίσης έχουμε ασχοληθεί με αρκετά θέματα που αφορούν τα λεγόμενα καινοτόμα τρόφιμα, τα novel food. Γι' αυτό κύριε Φαζέκας θα ακούσουμε την παρουσίασή σας και μετά θα σας θέσουμε ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Φαζέκας. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι μπορώ να προσέλθω στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή και να αναφέρω τα σχετικά με το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στην προστασία του περιβάλλοντος και τα συναφή περιβαλλοντικά θέματα. Εκ προημίου θέλω κάτι να θεωρήσω δεδομένο ότι για την Ουγγρική Προεδρία η προστασία του περιβάλλοντος και η αηφορία και στην περίοδο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς η Ουγγρική Προεδρία θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε εμείς τουλάχιστον να έχουμε εξίσου καλές, αν όχι καλύτερες, ε, ε, προϋποθέσεις διαβίωσης στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας σε σχέση με αυτές που βρήκαμε εμείς από τους γονείς μας. Οι αναβαθμισμένοι και μελλοντικέ ε, με, μελλοντικές θετικές προοπτικές περιβαλλοντική πολιτική δεν μπορεί να ε, διαχωριστεί από την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μόνο εκείνες οι χώρες και εκείνες οι περιφέρειες θα μπορούν να είναι επιτυχείς που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους ε, φυσικούς τους πόρους και θα προστατεύουν το περιβάλλον στο μέλλον μέγιστο βαθμό. Το μέλλον λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από αυτές τις κοινέ μας δράσεις και από την προσπάθειά μας ε, τις ευρωπαϊκές πολιτικές να τις προαγάγουμε όπως πρέπει και ενδιαφερόμαστε, έχουμε κάθε συμφέρον να είμαστε το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί συνεργαζόμενοι αναμεταξύ μας. Η Ουγγαρία θέλει πολύ στενά να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, για όλα τα θέματα. Θα επιθυμούσαμε να έχουμε μια Προεδρία που θα είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όσον αφορά το περιβάλλον έχουμε αρκετέ προτεραιότητε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω λόγο για τους υδάτινου πόρους, την πολιτική μας για τους υδάτινου πόρους. Η υδάτινοι πόροι είναι στρατηγική σημασία για τον 21ο αιώνα και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά και σίγουρα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ζήτημα και να ασχοληθούμε με την πολιτική για τους υδάτινους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αδύρυτη ανάγκη στην αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ, να λάβουμε υπόψη και την περιβαλλοντική συνιστόσα. Και κάτι άλλο. Πέρα από όλα αυτά, θα έχουμε και την βιοπικιλότητα που πρέπει να προστατευθεί και να προαχθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς. Έχουμε επίσης και το θέμα της ε, αντιμετώπισης ε, των ε, αποβλήτων και η στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να υποστηρίξουμε την μέγιστη, πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με την οδηγία Βέζο. Πρόκειται εδώ για τους κινδύνους που δημιουργούν τα απόβλητα όσον αφορά τη βιομηχανία. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το θέμα της συζήτησης για τον περιορισμό και την απαγόρευση της, ε, ε, και της διάδοσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Ουγγρική Προεδρία έχει δεσμευθεί ήδη και στοχεύει να αποσαφηνίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς διασκέψεις θα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα εδώ να επισέλθω στο θέμα που αφορά το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και την προκαταρκτική διάσκεψη του Ρίο και την 19η ε, ε, συνεδρίαση για την αηφορία στην ανάπτυξη, για την αηφόρο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό την συνάντηση των ε, όσων έχουν προσυπογράψει την συμφωνία του Όρχους και θα έχουμε και το θέμα των διαπραγματεύσεων για μια νέα στρατηγική για τον Ιδράργυρο και βλέπετε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ως Ουγγρική Προεδρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεξάρτητα από αυτό ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους για να επιτευχθούν αυτά τα σημαντικά, αυτή η σημαντική στόχη που έχουμε θέσει ενώπιόν μας. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να προαθούν όλα αυτά τα θέματα και είμαι εγώ πρόεδρος ε, της ε, προεδρεύω στο ε, Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και ξέρω ότι πρέπει να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά. Μόνο έτσι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και ε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε, με πιο εξειδικευμένο τρόπο στα θέματα. Όσον αφορά την αηφορία για την ε, χρήση των πόρων, ε, είναι αν, εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση και συνθήκη να είναι πιο σύγχρονη, πιο αηφόρος, πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη και η οικονομία της. Η Ουγγρική Προεδρία θέλει να συνεχίσει την πορεία που είχε ξεκινήσει και έδωσε, χάραξε η Βελγική Προεδρία και για τη στρατηγική 2020 με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα ισχύουν όλα αυτά πρέπει να τονίσω για την πρωτοβουλία αποτελεσματική στη χρήση των πόρων Ευρώπη η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων από πλευράς της Ευρώπης και να έχουμε ένα ε, οδικό χάρτη ακριβώς για να συνεχίσουμε αυτή μας την πορεία. Είναι ένα ευρύτατο φάσμα αυτό. Όσον αφορά την ε, αηφορία, όσον αφορά τα υλικά, τις, ε, τα απόβλητα, την ε, ανακύκλωση των αποβλήτων, την χρήση των υδάτινων πόρων, την καινοτομία. Ήδη τον Μάρτιο, σε σχέση με τις εργασίες του Συμβουλίου, θα έχουμε τις προτα... αναμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτά θα θέλαμε να πετύχουμε πέρα από αυτό στη συνάντηση του Συμβουλίου το Μάρτιο που προαναφέρθηκε να ε, υπάρξει πρόοδος. Η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί την αξιολόγηση του έκτου προγράμματος πλαισίου για το περιβάλλον ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση. Προσβλέπουμε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά. Η συζήτηση επ' αυτών των θεμάτων μπορεί να συνεισφέρει ώστε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον να μπορέσει να προετοιμαστεί και να καταρτιστεί και να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την αηφορία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις αναγκαίες στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Η βιοπικιλότητα εξακολουθεί να είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωσή της για μια νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα την έχει ε, δημοσιοποιήσει, θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις του Συμβουλίου. Στις 17 Ιουνίου θα διεξαχθεί ένα Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος. Σε αυτή την σύνοδο θέλουμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα τα οποία θα εγκρίνουμε για αυτά τα θέματα, για το περιβάλλον. Ευελπιστούμε ότι η ανακοίνωση έγκαιρα θα δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα αυτού του οδικού μας χάρτη. Είναι σημαντικό αυτή η στρατηγική μας από κοινού με την αλλιευτική πολιτική και την στρατηγική ε, που θα πρέπει να να ακολουθηθεί και για τη γεωργία και το περιβάλλον, να συνάδουν αυτά μεταξύ τους και για την δασοκομεία, δασοπονία, την αλληλεία, τη γεωργία και για τα ξένα προς τους ευρωπαϊκούς βιοτόπους ε, ε, φυτά ή ε, εκπροσώπους της πανίδας και χλωρίδας. Ε, η Ουγγρική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε το θέμα της ε, πρόσβασης ε, και της ίσης μεταχείρισης μετά τη συμφωνία της Ναγκόγια να διασφαλιστεί. Στόχος μας είναι κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011 να καταφέρουμε να πετύχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και η Ουγγαρία, αυτό το πρωτόκολλο να το, ε, έχουν, να το υπογράψουν. Μέσω αυτού έναντι των τρίτων χωρών θα αποστέλαμε ένα σημαντικό μήνυμα πόσο σημαντική θεωρούμε ότι είναι αυτή η νέα ρύθμιση αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελεστεί, διότι αυτό το πρωτόκολλο θα μπορέσει να αρχίσει να ισχύει μόνο όταν πρώτα ένα συγκεκριμένο αριθμό κρατών θα το έχουν προσυπογράψει. Μόνο τότε θα μπορεί να αρχίσει ε, μετά από αυτή την προϋπόθεση να εφαρμόζεται. Η υπογραφή λοιπόν η προσυπογραφή αυτού του πρωτοκόλου σε σχέση με τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών έχει τεράστια σημασία. Η Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το συμπληρωματικό πρωτόκολλο Κουάλα Λούμπουρ Ναγκόια να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε σχέση με την οικολογική ασφάλεια και το πρωτόκολλο της ε, Καρτα... Καρταγένης Καρθαγέλης, με συγχωρείτε. Όσον αφορά την, ε, τις διαπραγματεύσεις, ήδη το 2010 είχε υποβληθεί μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η πρόταση δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη σε σχέση με το ε, πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν για να περιορίσουν ή όχι τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Υπάρχουν διαφορές βέβαια. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να ξεκινήσουν και να προβούν σε έναν ανοιχτό ειλικρινή διάλογο αναμεταξύ τους. Όσον αφορά τις αβεβαιότητες όμως στο νομικό επίπεδο, αυτές θα πρέπει να έρθουν και να ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα πνοή στο έργο αυτό. Ο Επίτροπος Τζον Ντάλι υποσχέθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει, θα καταρτήσει ένα κατάλογο κατάλογο αιτίων και λόγων βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη την ε, ε, ένταξη των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα μπορούσαν να την περιορίσουν στην επικράτειά τους. Σε συνεργασία μαζί σας με το Ευρωκοινοβούλιο θα θέλαμε να επιτύχουμε σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα να επιτευχθεί νομική βεβαιότητα και νομική ασφάλεια η οποία την ομοφωνία που απαιτείται από πλευρά του Συμβουλίου σε σχέση με το, την προηγούμενη απόφαση του ε, Δεκεμβρίου 2008 θα διασφαλίζουν το νομικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι το σημερινό σύστημα διοδότησης όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να ξαναεξεταστεί και ενδεχόμενα να διαμορφωθεί σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Το θεωρούμε σημαντικό να εξεταστεί η αξιολόγηση των κινδύνων και μόνο έτσι θα μπορούσαν οι διοδοτούμενοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί υπό τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις και όρους να εξεταστούν σε σχέση με τους κινδύνους που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν όσον αφορά το περιβάλλον. Και μόνο τότε να μπορεί να δοθεί συνέχεια. Η πολιτική για τους υδάτινους πόρους έχει τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 θα εγκρίνει ένα έγγραφο για τη στρατηγική για τους υδάτινους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλείται blueprint, αποκαλείται δηλαδή σχέδιο ή πρότυπο και θα είναι ένα έγγραφο για τα κοινοτικά νομικά μέσα και πλαίσια για την πολιτική για τους ιδιάτινους, υδάτινους πόρους, για την αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων και θα υποβληθούν και προτάσεις για την βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύει αυτές τις διεργασίες και να τις ενδυναμώνει. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας θα καταλήξουμε σε έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτινων πόρων, για την πιο ολοκληρωμένη ε, αποδοτική ε, υδάτινη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και διαχείρισή τους θέλουμε ιδιαίτερη σπουδαιότητα να θέσουμε να πούμε ότι αναγνωρίζουμε στους εξής στόχους ακραίες ε, κλιματικές συνθήκες και μετεωρολογικά φαινόμενα και λειψιδρία και ανομβρία. Όλα αυτά τα ζητήματα τομεακά θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος αλλά και διατομεακά, διακλαδικά να δούμε ποιες, ε, ποιες ε, επιπτώσεις ε, προκαλούνται και να δούμε και τον ρόλο των υδάτινων πόρων και τον συνδυασμένο ρόλο οικοσυστημάτων, οικοβιοτόπων και υδάτινων πόρων. Θέλουμε επίσης να θέσουμε ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συνεργασία για τους υδάτινους πόρους μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η συνεργασία έχει, όπως προανέφερα, τεράστια σημασία αυτή η συνεργασία. Όσον αφορά την πράσινη ε, πολιτική, είναι σαφές ότι τα δύο θέματα, πολιτική για τη γεωργία και περιβάλλον, συναντώνται σε στενό βαθμό, ιδιαίτερα στενά. Οι ε, καλλιέργειες, ε, οι ε, δυνατότητες ε, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, βιοπικιλότητα, προστασία των εδαφών, προστασία των υδάτινων πόρων. Και όλα αυτά από πλευρά τους έχουν επιπτώσει στην αγροτική πολιτική. Η αηφορία απαιτεί από εμάς τους υδάτινους πόρους, να μην, τους ε, πόρους μας να μην τους εξαντλούμε. Πρέπει με αηφόρο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τους φυσικούς πόρους ε, και να τους διατηρούμε και να τους προστατεύουμε. Αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό ως προτεραιότητα για την ε, ε, αναδιάρθρωση και αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπως συζητείτε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ουγγρική Προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών Γερο... ε, ε Περιβάλλοντος έχει εγγράψει αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στη συνεδρίασή μας 15 Μαρτίου θα διεξαγάγουμε μια πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση και έτσι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στις διαπραγματεύσεις, πιο σημαντικές διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική μορφή και την κατεύθυνση της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθεί με τη συζήτηση αυτών των θεμάτων και θα τα προαγάγει αυτά τα θέματα και θα αντιδράσουμε τοποθετούμενοι στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουν να δούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι τα μέτρα για το περιβάλλον και για την αηφορία αλλά και για την προστασία του, της βιοπικιλότητας όλα αυτά θα συνεισφέρουν ώστε να πετύχουμε την αηφορία και την υλοποίηση των μέτρων για την ε, ε, κοινή αγροτική πολιτική. Δεσμεύεται η Ουγγρική Προεδρία για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να υποστηρίξει όλες εκείνες τις διαδικασίες και διεργασίες που θα οδηγήσουν σε μια απλούστευση της μορφής της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής και θα δώσουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν το δυνατόν περισσότεροι γεωργοί, ο μεγαλύτερος αριθμός ε, από πλευράς τους να αντιμετωπίσουμε την ε, μεταρρύθμιση της γεωργίας μειώνοντας τη γραφειοκρατική επιβάρυνση ε, στους γεωργούς και δημιουργώντας ένα πιο διαφανές πλαίσιο. Όσον αφορά τα απόβλητα από παλές ηλεκτρονικές συσκευές, ε, α, αυτά τα θέματα από μια οδηγία του 2002 διέπονται αυτή τη στιγμή. Αυτή η οδηγία που ε, το 2000, του 2008 πρέπει να ξαναεξεταστεί, να είναι πιο αποτελεσματική ώστε να έχουμε καλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση και να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Θέλουμε και σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πρόοδος. Έχει προχωρήσει η εργασία σε πολλούς τομείς, παρότι υπάρχουν, πρέπει να πω, διαφορές απόψεων σε κάποιους τομείς, όπως για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. Επίσης για την στοχοθέτηση όσον αφορά τη συλλογή αυτών των συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών που είναι πλέον απόβλητα και σε σχέση και με την ευθύνη των ίδιων των παραγωγών εταιριών που έχουν ε, δημιουργήσει και έχουν θέσει στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Θέλουμε επίσης ε, να δούμε και τις διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση κινητών ε, εξοπλισμών και μηχανών. Θέλουμε αυτό το θέμα να, τύχει, ε, να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Δεκέμβριο ξεκινήσαμε την οδηγία Σεβέζο ε, όπως την, σέβες όπως την αποκαλούμε για τα απόβλητα στον βιομηχανικό τομέα να την επανεξετάζουμε. Ξεκινήσαμε με αυτή την αναθεώρηση και ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Είμαστε ακράδαντα πεισμένοι ότι πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πυκνά κατοικημένη η Ευρώπη. Είναι μια βιομηχανική περιοχή, περιφέρεια, Ήπειρος και εδώ και αιώνες σημειώνεται αυτή η εξέλιξη και πρέπει να διασφαλίσουμε μια πορεία προς το μέλλον, μια μελλοντική πορεία που τις τιμές για το περιβάλλον, τις αξίες για το, του, ε, για το, του περιβάλλοντος θα τις διασφαλίζει ως αγαθά που θα δώσουμε, θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και που ε, αφορούν αυτή την πολιτική και που θα την ε, καταστήσουν εφικτή και μέσω της συνεργασίας. Χαίρομαι και προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία μαζί σας και προσβλέπω στο μέλλον. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ ε, ε, κύριε Προεδρεύον για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση του προγράμματός σας. Καλύψατε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι συμμετέχετε και στο Συμβούλιο Γεωργίας, διότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι πολυεπίπεδη, πολύπλευρη. Ενδιαφέρει και αυτή την Επιτροπή βεβαίως και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και ασφαλώς θα επανέλθουμε σε κάποια από τα θέματα τα οποία αναπτύξατε. επικοινότητα, παραδείγματο χάρη, πώς αυτή θα εφαρμοστεί. Ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα του στην Ευρώπη ε, πρόσβαση στα ωφέλη από τους γενετικούς πόρους. Και υπάρχει μία χώρα στον κόσμο που έχει ειδική νομοθεσία από αυτού και αυτή είναι η Νορβηγία. Οι Νορβηγοί έχουν ένα ABS δηλαδή νομοθεσία πρόσβασης και εποφελούς χρήσης, ε, ειδική νομοθεσία εδώ και τέσσερα χρόνια. Είναι λοιπόν προφανές ότι υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να σας υποβάλουν ερωτήσεις, διότι καλύψατε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, αλλά καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στην Οικονομική και Νομισματική Ενότητα της Κεντρικής Αφρικής και ο Πιέρ Νουγκουλού, πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, ε, επισκέπτεται την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας επισκέπτεστε. Ευρώπη και Αφρική έχουν στενές σχέσεις και επίσης αυτό το κοινοβούλιο έχει αναλάβει πολλές δεσμεύσεις έναντι αφρικανικών χωρών. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Επιστρέφω στα γερμανικά. Ε, έρχομαι λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών την πόρη. Ο Ρίτσαρτ Τζέιμπελ ε, ενθουσιάζεται με το θέμα αυτό, διότι είναι συντονιστής επί του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή και είπατε ότι έχει δύο πτυχές. Και ασφαλώς η υδάτινη πόρη, το νερό, είναι ε, μία από τις βασικές πτυχές. Και ε, πραγματικά χαίρομαι που έχω εδώ τον ειδικό υπουργό επί του θέματος και χαίρομαι ιδιαίτερος που η Ούγγροι είναι αποφασισμένοι να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στους υδάτινους πόρους κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους. Λοιπόν, έχουμε ε, γεωργούς οι οποίοι και ε, αγροτικέ αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, ε, στις οποίες το νερό διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη, την ευθύνη για τη διαχείριση των υδάτων. Μιλήσατε για τους υδάτινους πόρους, τις επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα και είπατε ότι θα υπάρξει μια ποιοτική προσέγγιση. Όπως γνωρίζετε, στην Νότια Ευρώπη αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη θα υπάρξουν, θα δημιουργηθούν προβλήματα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να διαθέτουμε επαρκείς ποσότητες ύδατος. Ασφαλώς υπάρχει η οικονομική πτυχή του ζητήματος και θα ήθελα να γνωρίζω τις οικονομικές επιπτώσεις. Η Ουγγρική Προεδρία έχει εντοπίσει τα ζητήματα και με απόλυτη λεπτομέρεια. Παραδείγματο χάρη, το θέμα του αφόδου πυρετού στην Ουγγαρία, τι επιπτώσεις είχε. Ο Πρόεδρος, θα έχουμε δύο γύρους ε, συζήτησης ο ένας γύρος σχετικά με το περιβάλλον και ήδη αναφερθήκαμε στο νερό και το δεύτερο κύκλος είναι η ασφάλεια τροφίμων. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ συγκεντρώστε τις ερωτήσεις θεματικά και ο Τάμπιτζ είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Ουγγρική Προεδρία σε στρατηγική σημασία θέματα όπως του υδάτινου πόρους δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα και το ανέφερε ο κ. Ζέμπερ πιο πριν. Έχουμε λήψη ιδρία, έχουμε διάφορα προβλήματα και, ε, που αφορούν όχι μόνο την λεκάνη της Μεσογείου και τις χώρες γύρω από αυτήν, αλλά και αφορούν για παράδειγμα και την λεκάνη του Δούναβη και τις ε, όμορε χώρες. Η ερώτησή μου αφορά και εντοπίζεται σε αυτό το θέμα εν μέρη εσείς ε, ως ε, Προεδρεύων Υπουργό, ε, αρμόδιο για την γεωργία, του διάτρου πόρου και την ανάπτυξη τη υπαίθρου, ποιε πρωτοβουλίε θα αναλάβετε στο Συμβούλιο Υπουργών για όλα αυτά τα θέματα. Από την άλλη πλευρά, Μόλις τώρα ξεκινά αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα, το δεύτερο σημαντικότερο πρόγραμμα για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική για τον Δούναβη. 12 χώρες εμπλέκονται, 8 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη στρατηγική για τον Δούναβη απορρέει το πρόβλημα κατά πόσον ο Δούναβης θα είναι ανοιχτό στην αυσιπλοεία ή όχι και κατά πρώτο λόγο βέβαια στο νότιο τμήμα του Δούναβη Πώς θα μπορούσε η ναυσιπλοεία στον Δούναβη να ενδυναμωθεί και να επεκταθεί, να υποστηριχθεί αυτό το εγχείρημα. Αυτό θα ήταν αφενός πολύ καλό για τη γεωργία και αφετέρου έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και γι' αυτό πρέπει το περιβάλλον να προστατευτεί ιδεόντως. Πώς θα μπορούσαν αυτές οι αντιφατικές πλευρές να συγκεραστούν και να εναρμονιστούν μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκέρνιαν μπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό Φαζέκας για την παρουσία του εδώ και για την παρουσίαση του προγράμματος του που είναι πολύ πιο φιλόδοξο από ότι στην γραπτή μορφή διότι εγώ το διάβασα και αυτό είναι πράγματι πολύ θετικό και ελπίζω ότι αυτή η προσωπική δέσμευση θα ε, πάρει σάρκα και οστά τους προσεχής ε, μήνες. Βιοπικιλότητα. Για μένα το 2010 ήταν ένα έτος υποσχέσεων με κορύφωση στη διάσκεψη κορυφή της Ναγκόγια όπου ως διεθνής κοινότητα αναλάβαμε δεσμεύσεις. Ενώ το 2011 θα πρέπει να είναι η έναρξη της δράσης των ενεργειών. Διότι ακούσαμε πάρα πολλές υποσχέσεις εδώ και δέκα χρόνια ε, σχετικά με την βιοπικιλότητα. Είναι λοιπόν θετικό που θέλετε να συνδυάσετε την βιοπικιλότητα με την κοινή αγροτική πολιτική, την πολιτική αλληλείας και επιδιώκετε να επικυρωθεί το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Το ερώτημά μου λοιπόν συνδέεται με το άλλο έγγραφο της Ναγκόγια, το της στρατηγικής. Ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα προσεχή 10 χρόνια είναι οι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις που συνδέονται με την βιοπικιλότητα. Τι, πώς λοιπόν θα ξεκινήσετε αυτό το έτος δράσης στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό που είναι μαζί μας σήμερα. Χαίρομαι γιατί υπογραμμίσατε ένα θέμα το πολύ σημαντικό και στρατηγικό θέμα των υδάτινων πόρων. Είναι κάτι το οποίο αφορά επίσης και την, νομοθεσία των, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ξέρετε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι στην Ουγγαρία το προηγούμενο φθινόπωρο με την ε, ερυθρά λάσπη, την κόκκινη λάσπη από τη μονάδα αυτή επεξεργασίας. Επισκέφτηκα την περιοχή και συναντήθηκα τότε και με τον τότε υφυπουργό υπεύθυνο για τα θέματα αυτά που είναι ανάμεσά μας σήμερα. Είχαμε αλληλογραφία επίσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από το συγκεκριμένο πρόβλημα και από ό,τι φάνηκε η ερμηνεία την οποία δίνει η Ουγγρική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία είναι κάτι το οποίο δημιουργεί παρανοήσεις σε δύο τουλάχιστον θέματα. Πρώτο, η οδηγία, η αρμόδια για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, τις εξορρυκτικές, η Ουγγρική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή της. Εάν όμως είναι εφαρμόσιμη η συγκεκριμένη οδηγία για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες, θα έπρεπε να έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Το δεύτερο θέμα στο οποίο υπάρχει διαφορά από πλευράς της Επιτροπής, μεταξύ της Επιτροπής και του Ουγγρικής Κυβέρνησης, αν αυτή η κόκκινη λάσπη που προέρχεται από την εξόριξη υλικού για αλουμίνιο, σε ποια κατηγορία ανήκει. Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα έπρεπε, επειδή ακριβώς ε, είναι είναι υλικό το οποίο προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα θα έπρεπε να χαρακτηριστεί σαν επικίνδυνο υλικό και να μπει στην αρμόδια κατηγορία. Αλλά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν η Ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε πού θα ταξινομήσει τη συγκεκριμένο υλικό και αν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η θέση ε, της Ουγγρικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ε, περιοχών που έχουν μολυνθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες δεν ασχολούνται καθόλου με την αποκατάσταση συγκεκριμένων περιοχών, ε, ιδιαίτερα από χημικές ουσίες. Υπάρχουν ε, πολλά παραδείγματα στη δική μου χώρα σαν παράδειγμα όπου ε, έχουν ε, αποθηκευθεί σε υπόγεια σε αποθήκες πάρα πολλές χημικές ουσίες. Υπάρχουν, υπάρχει περιεκτικότητα χρωμίου σε ορισμένους υδάτινους πόρους της χώρας μου 8 φορές περισσότερο από το επιτρεπόμενο χρησιμοποιούνται τα ύδατα αυτά για την, ε, για την παροχή νερού στα ζώα σαν παράδειγμα και στην κτηνοτροφία και ε, υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν από όλες αυτές τις ουσίες. Υπάρχουν εν πάση περιπτώσει 70 τέτοιες επικίνδυνες ουσίες από τις οποίες το χρώμιο είναι η πιο επικίνδυνη και η πιο γνωστή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Σκοπεύετε εσείς να προχωρήσετε ακριβώς ε, την οδηγία αυτή έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις για όλες τις χώρες έτσι ώστε κάποιες περιοχές που έχουν μολυνθεί να αποκατασταθούν άμεσα γιατί αλλιώς θα δημιουργήσουμε πάρα πολλά προβλήματα ε, και στη φύση γενικότερα και στους ανθρώπους ε, οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και που αποδεικνύεται και από τον αριθμό των πολλών ερωτήσεων προς την Ουγγρική Προεδρία και σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας της. Τώρα, όσον αφορά την διαχείριση των υδάτινων πόρων και όσον αφορά και την βιολογική διατήρηση της βιοπικιλότητας υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις που επικεντρώνονται πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να αναφέρω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα εργασίας, στο οποίο εμπεριέχεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα το θέμα των υδάτινων πόρων κατά το επόμενο διάστημα. Είναι δυνατόν όμως κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου να μην μπορεί η Ουγγρική Προεδρία να επιτύχει την έγκριση ενός νομοθετικού προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το 2012 να αναθεωρήσει τα μέχρι σήμερα ενισχύει νομικά μέσα και πλαίσια όσον αφορά και την ε, εφαρμογή τους, πρώτα απ' όλα την οδηγία για το νερό. Και τις διαφορετικές δυνατότητες και διατάξεις που συνδέονται με τη διαχείριση του νερού, ώστε μέσα στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών να μπορέσουν να επανεξεταστούν. Το 2012 θα υποβάλει ένα έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σφαιρική στρατηγική για το νερό, ένα blueprint όπως το αποκαλούμε και θα υποβάλει έτσι προτάσεις για μια μελλοντική νομοθετική ρύθμιση αυτών των συνιστοσών στο μέλλον. Η Ουγγρική Προεδρία θα ήθελε στον τομέα της διαχείρισης του νερού πρώτα απ' όλα αυτή η διεργασία να προαχθεί, ώστε οι, διάφορες, οι διάφοροι τομείς να μπορέσουν να συγκλίνουν. Θέλουμε να μπορέσει να υπάρξει έγκριση από πλάσου του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτινων πόρων για την αηφορία της πολιτικής για τους υδάτινους πόλους τον Ιούνιο θέλουμε προτιθέμεθα να εγκρίνουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Πέρα από αυτό είναι σημαντικό να δούμε ότι η οδηγία, η οδηγία για την ποιότητα του νερού θα μπορεί να στήχει εξέτασης, ε, περαιτέρω εξέτασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό σε αυτό το επίπεδο κατά τους επόμενους έξι μήνες ε, να πούμε ότι αυτό θα είναι το κυριότερο έργο μας. Όσον αφορά τις τοξικές ουσίες ε, στο νερό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει να, ε, την επανεξέταση της ε, οδηγίας αυτής και ελπίζουμε ότι στο επόμενο έγγραφο που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμπεριέχονται οι αντίστοιχες προτάσεις. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να δρομολογήσουμε διαφορετικά, διαφορετικές πρωτοβουλίες για τους υδάτινους πόρους και να συνδεθούν αυτά με το blueprint της Επιτροπής και προσβλέπει η, Ευρωπα... η, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευρά της Ουγγαρίας σε προόδους που θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Ορέστε Ρώση, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα σχέδια ή προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτού του εξειδικευμένου προβλήματος. Θεωρούμε όμως ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλη σημασία, διότι η προστασία των ε, νερών είναι σημαντικότατο θέμα για την Ευρώπη όσον αφορά την βιοπικιλότητα και εδώ υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις που διατυπώθηκαν για αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι θα προσυπογραφεί το πρωτόκολλο της Ναγόγια και έτσι η Ουγγρική Προεδρία θα πρέπει να προετοιμάσει μια κοινή θέση που θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Ιούνιο 2011 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτησή μας αυτή και θέλουμε σε άτυπες συνεδριάσεις πραγματογνωμόνων να ε, συνοδευτεί αυτό το έργο και να το παρακολουθήσουμε ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Και με βάση αυτό το, αυτή την κοινή θέση θα καταλήξουμε στην έκτη διακυβερνητική διάσκεψη και όσον αφορά θέματα χρηματοδότησης, θα ήθελα να σας πω ότι η Ουγγρική Προεδρία ακολουθεί μια στρατηγική για την κινητοποίηση ε, κονδυλίων και χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Θέλει να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και σε συνέχεια συνεργαζόμενοι με τις προτάσεις της ε, ε, Βελγικής Προεδρίας θα υπάρξει ένα έγγραφο το οποίο ε, βρίσκεται υπό που θα εξετάζει τη στρατηγική, θα διατυπώνει τις επιμέρους τομεακές στρατηγικές που θα μπορούν να συγκλίνουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεμάτων Εντάσσεται επίσης ότι στην χθεσινή ακρόαση του κυρίου Ποτοτσνίκ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για την αποδοτικότητα ε, και αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων. Αυτή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σίγουρα αποτελεί μια πρόοδο. Όλες οι νομικές διατάξεις ε, θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν ώστε η αηφορία να διασφαλιστεί και να υπάρξει η υποστήριξη σε σχέση και με το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τη στρατηγική τώρα για τον Δούναβη, μια άλλη πτυχή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η στρατηγική για τον ποταμό Δούναβη έχει τεράστια σημασία ως πρωτοβουλία για όλες τις όμορες χώρες ε, που ε, βρίσκονται ε, αμφωτέρωθεν του Δούναβη. Μπορεί να αποτελέσει και θεμέλιο για μια συνεκτική, συναφή πολιτική ως προσέγγιση για άλλες περιφέρειες. Τα κονδύλια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια εναρμονισμένη προσέγγιση και έτσι μπορούμε να, να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλύτερο, σε ένα πολύ πιο βελτιωμένο αποτέλεσμα για την, κοινωνική, για την περιφερειακή συνοχή και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Είναι πολύ σημαντικό με συνεκτικό τρόπο να διαμορφωθεί αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες χώρες και οι χώρες αυτές να καταφέρουν στο τέλος τέλος να αποκτήσουν να συμμετάσχουν εθελοντικά ε, σε αυτό το πρόγραμμα. Ήδη υπάρχει ε, επιτυχής ε, συνεργασία που έχει αναπτυχθεί και διαμορφώνεται. Παράδειγμα, η Συμφωνία για τα Καρπάθια, το Φόρουμ για τον ποταμό Τίσα, επίσης η Επιτροπή για τον Δούναβη. Θεωρούμε τούτων λεχθέντων συνολικά ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική για τον Δούναβη κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας θα πρέπει να μπορέσουν να εγκριθούν και είμαστε έτσι πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας κύριοι Ευρωβουλευτές γιατί ο συντονισμός είναι πολύ σημαντική υπόθεση για αυτούς τους στόχους. Πολλά ερωτήματα τίθενται, ζητήματα τίθενται σε σχέση με το θέμα κατά πόσον η ναυτιλιακή ανάπτυξη, στο, οι ναυτιλιακές μεταφορές ε, θα μπορέσουν να ε, επεκταθούν στο Δούναβι έχουν ε, υπάρχει ένα σύνολο ε, θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν και συμφωνούμε πιστεύω ότι αν θέλουμε και όταν θέλουμε να προαγάγουμε την κινητικότητα θα πρέπει να εξευρεθούν πάντα να εξευρίσκονται λύσεις που θα σέβονται το περιβάλλον και θα το προστατεύουν. Φυσικά η ναυσιπλοεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να υποστηριχθεί η ναυσιπλοεία στον η Δούναβη. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να συνάδουν με την οδηγία για το νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την νατούρα Natura 2000, την προστασία της φύσης 2000 και τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις και ρήτρες που διέπουν αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι όταν κάνουμε λόγο για ναυσιπλοεία θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και να βλέπουμε ότι η ναυσιπλοεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στον ποταμό και τις προϋποθέσεις που προσφέρει και όχι ο ποταμός να προσαρμόζεται εκείνος στις ανάγκες του με την διευρυμένη ναυσιπλοεία. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα δασοκομικά θέματα υπήρξαν αρκετά ερωτήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αναφέρατε αυτή την πτυχή, διότι τα δασοκομικά θέματα δεν είναι μόνο και όσον αφορά και τη δασοπονία σημαντικότατα όσον αφορά την ε, ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ισχύουν βέβαια οι εθνικές ε, πολιτικές και ρυθμίσεις, αλλά είναι αμφίδρομη η επίδρασή τους όσον αφορά για παράδειγμα την υπερθέρμανση του πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές καθιστούν αδύρυτη ανάγκη να ασχοληθούμε με τα δάση μας. Στην Ουγγαρία έχουμε 2 εκατομμύρια εκτάρια δασικών εκτάσεων, δασών. Στο παρελθόν ήταν πολύ μεγαλύτερη η έκταση που καλυπτόταν από τα δάση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναφέρουμε ότι η αναδάσωση έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα και σπουδαιότητα για αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πράσινη βίβλο καλύπτοντας αυτά τα θέματα αναμένουμε και προσβλέπουμε ότι η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποβληθεί το Μάρτιο. Με βάση αυτή την ε, γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, επ' αυτών των θεμάτων. Αναφέρθηκε επίσης το πρόβλημα των ε, υλικών που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές και όσον αφορά και τις εκπομπές ρήπων, διότι φυσικά εδώ το ξύλο, τα δάση, το, απορροφούν εκπομπές ρήπων διοξίδιο του άνθρακα και όταν έχουμε αποψήλωση των δασών για να χρησιμοποιείται το ξύλο ως οικοδομικό υλικό τότε δημιουργούνται προβλήματα με την δυνατότητα απορρόφησης ε, και αφομοίωσης του διοξιδιού του άνθρακα από τα δάση. Θα διεξαχθεί μια διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη και θα έχουμε μια νομοθετική ας το πω έτσι πρόταση που θα προετοιμαστεί για την, για την προστασία των δασών. Δεν γνωρίζουμε αν θα καταφέρουμε ε, όλες τις ε, προθεσμίες, αλλά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Τέθηκε ένα ερώτημα για τον αυθόδη πυρετό στη Βουλγαρία και είμαι πισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στη διάθεσή της τις αναγκαίες ε, θεσμικές ε, και διοργανωτικές δομές ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα όπως ε, θα έπρεπε. Από πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας έχουμε προβεί σε ε, παρασκευή των ε, προετοιμασία των αναγκαίων συζητήσεων. Στις 18 Ιανουαρίου ήδη διεξήχθη μια πρώτη συνεδρίαση από πλευράς των ε, ανώτατων υγειονομικά και κτηνιατρικά υπεύθυνων. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ομάδα πραγματογνωμόνων θα αποσταλεί στη Βουλγαρία ώστε να εξεταστούν τα γεγονότα αυτής της αυθόδους, ας το πω αυτού του αυθόδους πυρετού περιοχή του ποταμού Τίσα και τα συναφή θέματα εντάσσονται και συνδέονται και με την πολιτική για τον Δούναβη. Υπάρχει όμως εδώ ένα κλιματικό φαινόμενο το οποίο α, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα όσον αφορά και την ε, ξηρασία ή και την λειψιδρία ε, εκάστοτε. Είναι ένα πρόβλημα ότι έχει σημειωθεί έλλειψη υδάτινων πόρων, δηλαδή η σημαντική ανομβρία και μέσω αυτής ε, ε, προβλήματα ξηρασίας, ε, υπάρχει κινητοποίηση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν προγράμματα ώστε το επίπεδο, η στάθμη των υδάτων στις λίμνες να μπορέσει να βελτιωθεί, να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ένα νέο πρόγραμμα από πλευράς Ουγγαρίας ε, που αποκαλείται βαρσαρ Hey πρόγραμμα. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ε, εργαζόμαστε σφαιρικά για να αντιμετωπιστούν όλα τα αίτια. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σίγουρα κυρίες και κύριοι. Μία περαιτέρω ερώτηση που απευθύνθηκε ήταν το θέμα σε σχέση με την ε, κόκκινη λάσπη και την ε, ε, καταστροφή αυτή που έπληξε την Ουγγαρία. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ε, θέμα και γι' αυτό δεν μπορώ να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες βέβαια. Ωστόσο η Ουγγαρία ανέλαβε την, ε, τα αναγκαία μέτρα ε, πάντα που συνάδουν πάντα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την οδηγία για τα απόβλητα που εγκρίθηκε το 2008 και που αναφέρει ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία αποβλήτων η κόκκινη λάσπη. Στη συνέχεια όμως διορθώθηκε αυτή η έλλειψη και προβλέπεται φαίνεται πλέον τώρα ότι ένα υποπροϊόν αυτής της βιομηχανίας αλουμινίου είναι αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίζεται μέσα στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφεξής αυτό θα ισχύει ε, και στην Ουγγαρία φυσικά. Αυτό θα σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές παραγωγής αλουμινίου θα εποπτεύονται πλέον από τις Ουγγρικές αρχές και δεν θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει επανάληψη ε, αυτού του συμβάντος στο, μέλλον. Υπάρχει και το θέμα της αδειοδότησης σε σχέση με αυτό το πλαίσιο, την καταστροφή αυτή που ε, είχαμε. Η τεχνολογία έχει πλέον αλλάξει, η μέθοδος που χρησιμοποιείται από αυτή τη μονάδα έχει πλέον τροποποιηθεί και δεν χρησιμοποιείται η παλαιά μέθοδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Τρεις έχουν ζητήσει ε, το λόγο για περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα ήθελα να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα για να περάσουμε μετά στη συζήτηση σε θέματα υγείας. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν ε, ε, σχετικά με το περιβάλλον. Έτσι, η κυρία Κλάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Προεδρεύον, σχολιάσατε την ε, μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ. Δεν είναι θέμα που ενδιαφέρει άμεσα αυτή την Επιτροπή. Αναφερθήκατε όμως στις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι δεν είστε ικανοποιημένος με τις προτάσεις του Επιτρόπου Ζέλλας και ιδιαίτερα όσον αφορά στα κίνητρα για φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες. Ωστόσο το ερώτημά μου ουσιαστικά αφορά τη στρατηγική ε, επί των πρώτων υλών. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τον ρόλο ε, το ρόλο που θέλετε να δώσετε στα ανανεώς, στις ανανεώσιμες πρώτες ε, ύλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα αυτό το οποίο πηγαίνει στην δεξαμενή των οχημάτων. Σχετικά τώρα με την Σχετικά με τα βιοαέρια, θα ήθελα να μάθω ποια είναι η θέση σας ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχω ένα σύντομο ερώτημα. Είμαι ευγνώμων που αναφερθήκατε στα γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το ερώτημά μου έχει ως εξής η Κομισιόν ε, πρόκειται να δημοσιεύσει έναν κατάλογο. Πιστεύετε ότι η τάση είναι να έχουμε έναν ευρωπαϊκό κατάλογο για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή ε, μήπως υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο ε, Συμβουλίου να διευθετηθεί το ζήτημα. Και τώρα αυτό το ερώτημα μπορείτε να θέσετε στο δεύτερο μέρος όταν θα συζητήσουμε τα θέματα υγείας. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να απαντήσετε ε, στην ερώτηση αυτή στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης που θα αναφερθούμε σε θέματα υγείας. Σας παρακαλώ πολύ να συγκεντρώσουμε τα θέματα, διαφορετικά θα εμπλακούμε. Ο κύριος ε, έχει την τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω το εξή ερώτημα. Προτίθεστε να Ολοκληρώστε τις διαπραγματεύσεις ε, για τα απόβλητα από ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικούς ε, ε, ηλεκτρονικές συσκευές. Και αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε να απαντήσετε στην ερώτηση. Έχω μία ερώτηση σχετικά με το αέριο. Ε, σχετικά με τα αέρια από ε, σχιστόλυτο και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, έχουμε μία διαφορά με τις Ηνωμένε Πολιτείε γιατί τούτο ε, ρηπαίνει τον υδάτινο ορίζοντα και επηρεάζει το πόσιμο νερό. Θα ήθελα να μάθω κύριε Υπουργέ, εάν είστε υπέρ μιας ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με αυτό τα αέρια από σκιστόλουδο, ούτως ώστε να αναπτύσσεται τεχνολογία η οποία δεν ρηπαίνει τον υδάτινο ορίζοντα και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη χρησιμοποίηση ε, αυτών των αερίων από σκιστόλιθο. Έχετε το λόγο να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Ε, θέλουμε να έχουμε χρόνο και για να απαντήσετε στα ερωτήματα σχετικά με την υγεία, κύριε Υπουργέ. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω σύντομα να αποφασίσω παρότι αυτά τα θέματα δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα δική μου. Όπω και οι συνάδελφοί μου στο Ουγγρικό Υπουργείο, θα ήθελα να υπάρξει η δυνατότητα αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να υπησέθω σε ερωτήσεις και να απαντήσω, γραπτός να δοθούν απαντήσεις ή να έρθω σε διαβούλευση μαζί σας. Όσον αφορά την πράσινη αγροτική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει σχεδιάσει έτσι ώστε οι άμεσες, η ε, άμεση υποστήριξη να έχουν μια συμπληρωματική συνιστόσα που θα αποκαλείται πράσινη συνιστόσα. Αυτό υφίσταται και στο σημερινό σύστημα σε κάποιο βαθμό. Όμως θα υπάρξει μεγαλύτερο πλαίσιο υποστήριξης όταν θα ανταποκρίνονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε αυτό το πρασίνισμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και συνάδει με τις αρχές που προηγούμενα εξετέθησαν. Είναι πολύ σημαντικό θεωρώ οι απόψεις από των κρατών μελών να συλλεγούν και να καταγραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Η Ουγγρική Προεδρία ε, θα ε, στοχεύει σε, ένα πρώτο, σε μια πρώτη φάση να υπάρξουν συμπεράσματα από πλευρά του Συμβουλίου Συμβουλίου επ' αυτών των προτάσεων. Διάφορες οργανώσεις και σύλλογοι γεωργών, διάφορα κράτη-μέλη έχουν ήδη πει ότι καλό θα ήταν αν θα ήταν δυνατόν οι μεταβολές, οι τροποποιήσεις ε, όσον αφορά τους κανονισμούς να είναι αποτελεσματικές, στοχοθετημένες και το σύστημα ενισχύσεων ε, ε, επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην δυσχερανθεί ε, περισσότερο, ε, να μην κατασταθεί πιο περίπλοκο, να είναι πιο απλό και λειτουργικό. Όλοι συμφωνούν συμφωνούν να είναι πιο απλό και πιο εύκολα να μπορεί κανείς να προσαρμοστεί σε αυτές τις ρυθμίσεις σε σχέση με το πρασίνισμα της γεωργικής πολιτικής. Υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία, ήδη κάποια στοιχεία σε αυτό το, σύστημα τα οποία λειτουργούν με πολύ θετικό τρόπο και που καταδεικνύουν ότι στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια φιλική προς το περιβάλλον γεωργία έχει τεράστια σημασία. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την αποδοτικότητα των πόρων και την αηφορία. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι, και το τονίζω αυτό, ότι η αηφορία όσον αφορά την διαχείριση και την εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Εμείς ε, τους φυσικούς πόρους και την εκμετάλλευσή τους πρέπει να τη σχεδιάσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η περιβαλλοντική πολιτική που θα βασίζεται στην ανοιχτή οικονομία της αγοράς θα μπορεί να είναι κινητή κινητήρια μηχανή, κινητήρας ε, για την ανάπτυξη και την δημιουργία απασχόλησης. Πρέπει να τεθούν τα θεμέλια ώστε να υπάρξει καινοτομία που θα μπορέσει να δράσει και να συνοδεύει αυτές τις πρωτοβουλίες. Και το περιβάλλον να αποκομίσει κέρδος αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα τονωθούν στην απασχόληση. Όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας, θα πρέπει γι' αυτό τον λόγο να μπορέσουν να προβλέπονται και να σχεδιάζονται έτσι ώστε η αηφορία των πόρων να είναι πάντα στο επίκεντρο. Και δεν έχει κανένα νόημα να διαφοροποιούμε τα πράγματα μεταξύ καλών εντό εισαγωγικών και κακών βιομηχανικών τομέων όλοι οι τομείς, οι βιομηχανικοί τομείς θα μπορούν με αηφορία να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν. Οι στοχοθετημένες λοιπόν επενδύσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε πιο φιλοπεριβαλλοντικά να μπορέσουν να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν αυτοί οι βιομηχανικοί τομείς. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την επίτευξη των στόχων μας όπως τους προανέφερα όσον αφορά το βιοαέριο και τα βιοκαύσιμα. Και εξάλλου τις δυνατότητες παραγωγής τους. Είναι ένα πολύ, πολύ περιπλοκό θέμα αυτό και δεν έχουμε επαρκή χρόνο που να για να μπορέσουμε να το καλύψουμε. Υπάρχουν όμως ε, απόβλητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ε, ε, ενδυνάμωση αυτού του τομέα και δυνατότητες που θα δώσουν ένα πιο θετικό απολογισμό στο τέλος ε, των ενεργειακών πόρων. Είμαι πεισμένος ότι η καινοτομία και η έρευνα όσον αφορά την τεχνολογία θα δώσουν νέες δυνατότητες που θα είναι πολύ, νέες εναλλακτικές λύσεις που θα είναι πολύ αποτελεσματικές. Υπήρξε επιπλέον ακόμα μια ερώτηση που αφορούσε την οδηγία, την ε, ε, και πρέπει εδώ να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντική η υπόθεση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Θα θέλαμε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα που εκκρεμούν ακόμη και θα θέλαμε πάντα να, συνεργαζόμαστε μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εξέβρεση λύσεων. Θα περάσουμε στα θέματα της υγείας, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν αρκετά θέματα που τέθηκαν και γι' αυτό θα ήθελα να είστε πιο σύντομοι σε ερωτήσεις σας για να έχει ο Υπουργός χρόνο απάντησης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς για τη διοξίνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Είχε τεθεί θέμα και με τις πιθανές απαγορεύσεις εισαγωγών προϊόντων. Τίθεται επίσης το θέμα των ελέγχων και των μέσων ελέγχου που έχουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τη διοξίνη. Ένα άλλο τομέα είναι τα λεγόμενα καινοτόμα τρόφιμα, τα novel foods. Εδώ έχουν αποτύχει οι προσπάθειες που έχουν κάνει διάφορες προεδρίες και σε σχέση με τους κλόνους και σε σχέση με τη δεύτερη γενιά. Υπάρχει πάντα η απαγόρευση βέβαια κλωνοποίησης. Νομικές ρυθμίσεις υπάρχουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει όμως να ελέγχεται το τι έχουν καταναλώσει τα ζώα και τι, ε, επίσης έχουν, τι προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί γενικότερα στην ανατροφή των ζώων. Για την κλωνοποίηση είναι πιο εύκολος ο έλεγχος αρκεί να γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο πατέρας και ποια η μητέρα του συγκεκριμένου ζώου. Και σε σχέση με την ετικετοθεσία των τροφίμων ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάπου θα καταλήξει αυτή η ιστορία και θα συμφωνήσουμε. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι σαν παράδειγμα από τις ετικέτες που τίθενται στις απομιμήσεις. Ντάγμα. Ήμουν παρούσα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των προγραμμάτων γενικά και από πλευρά της Ουγγρικής Προεδρίας πάντα παίζουν με τη φράση που λέγει προστασία του καταναλωτή. Αυτό τουλάχιστον γινόταν μέχρι τώρα. Εσείς είστε υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας τροφίμων λοιπόν κύριε Υπουργέ. Περιοριστήκατε βέβαια στο να αναφερθείτε στο χαρτοφυλάκιό σας, σας ε, λέγοντας ότι είναι πολιτική περιβάλλοντος γενικά και δεν αναφερθήκατε συγκεκριμένα στα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων. Γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Τι θα γίνει με τα καινοτόμα τρόφιμα σαν παράδειγμα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Θα έπρεπε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε τη στήριξή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την κλωνοποίηση των ζών, για την απαγόρευση της κλωνοποίησης των ζών, όπως επίσης και για, την λεγόμενη, για τα διάφορα επίπεδα ψήξης. Αναφερθήκατε πάρα πολύ, συχνά, πάρα πολύ συνοπτικά στα γενετικά τροποποιημένα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Απαιτείται να υπάρξει μια λύση η οποία να είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει και εδώ να συνεργαστούμε και να ζητήσετε και εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει με τη σειρά της από την ε, αρμόδια υπηρεσία να λάβει υπόψη την κοινοτική νομοθεσία πλήρως. Πρέπει λοιπόν η υπηρεσία αυτή στην Πάρμα της Ιταλίας να εφαρμόζει σωστά την κοινοτική νομοθεσία. τι γίνεται με την αδειοδότηση κυκλοφορίας ζωοτροφών σαν παράδειγμα. Θυμάστε τι είχε γίνει με την κρίση της τρελής αγελάδας. Δεν θα πρέπει να ξανσυμβεί κάτι τέτοιο. Και τι θα γίνει και με τις ετικέτες ε, στις ζωοτροφές. Έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία του σχεδίου για τη δεύτερη ανάγνωση. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συμφωνία. Θα πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει και με τις απομιμήσεις. Λοιπόν κύριε Υπουργέ θα σας δώσω σε λίγο το λόγο γιατί πρώτη πριν απαντήσετε θα κάνετε μια εισαγωγική παρουσίαση. να συνεχίσω λίγο αυτά τα οποία είπε η Ροντ Μπέρεντ. Θέλω να συμπληρώσω κατά κάποιο τρόπο τις ερωτήσεις της. Εγώ είμαι η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα γενετικά τροποποιημένα. Δεν ήθελα να σας μιλήσω όμως για τη συγκεκριμένη πρόταση. Ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία αυτών που είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Για τα γενετικά τροποποιημένα το βασικό θέμα είναι να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία του 2008. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος του 2008 για την αξιολόγηση των κινδύνων. Η ΕΦΣΑ δεν εφαρμόζει αυτά που ζήτησε το Συμβούλιο του 2008 δεν αναγνωρίζει τις επιστημονικές δοκιμές και πειράματα, δεν λαμβάνει υπόψη ε, στην αξιολόγηση των κινδύνων μακροπρόθεσμα. Δύο νέες διατυπώσεις των κατευθυντηρίων γραμμών προτάθηκαν, η μία αφορά την υγεία και η άλλη το περιβάλλον. Τα έγγραφα αυτά συνεισφέρουν. Από την άλλη όμως ε, έχουν και κάποιες αδυναμίες και κάπου υπαναχωρούν σε σχέση με τις υπάρχουσες πρακτικές. Είναι σημαντικά τα έγγραφα αυτά βέβαια, για τα συμπεράσματα του 2008. Διαρωτώ με λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσετε σε επίπεδο συμβουλίου, γιατί θα πρέπει να συνοδεύουν όλες τις συζητήσεις για τη νέα οδηγία. Θα συζητήσετε επίσης το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο κύριος Ντάλι, ο Επίτροπος Ντάλι, μας είπε εδώ και λίγες μέρες ότι θα κάνει προτάσεις συγκεκριμένες. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη πολλές ερωτήσεις ε, διατυπώθηκαν και χαίρομαι φυσικά για αυτό το γεγονός. Όμως ήδη έκανα λόγο με τον κύριο Πρόεδρο προηγούμενα ότι θα έχω ξεχωριστή δυνατότητα που θα μου δοθεί να παρέμβω για την ασφάλεια τροφίμων. Και έτσι με τον κύριο Πρόεδρο έχοντας αυτά συζητήσει. Γι' αυτό δεν έκανα λόγο για αυτά τα θέματα μέχρι τώρα. Είναι αυτονόητο φυσικά ότι υπάρχουν θέματα που και αμφότερα και στις δύο πλευρές ε, ε, παρουσιάζονται και τίθενται και στην πρώτη παρέμβαση και στη δεύτερη. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η νέα ε, ρύθμιση θα έχει προτεραιότητα από πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας. Είμαι πεισμένος ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη αξία για αναβαθμισμένα και πολύ καλής ποιότητας ε, τρόφιμα και με πλήρη πληροφόρηση. Και όταν θέλουν να αγοράζουν οι καταναλωτές συμφωνούμε ότι θέλουν να γνωρίζουν τι βρίσκεται πίσω από τη συσκευασία, μέσα στη συσκευασία ως προϊόν. Θέλουμε λοιπόν διεξοδικά να πληροφορούνται για το προϊόν το οποίο τους προσφέρεται προς αγορά. Η παραγωγή τροφίμων μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής τροφίμων, μέσα από τις νέες τεχνολογίες, έχουμε και νέες ουσίες και νέες, νέες ουσίες που χρησιμοποιούνται μέσω παγκοσμιοποίησης και εντάσσονται στις μεθόδους παραγωγής και ε, παρασκευής των τροφίμων Υπάρχει όμως, ε, δεν υπάρχει και τέτοια εμπιστοσύνη σε όλα αυτά και υπάρχουν αβεβαιότητες και ανασφάλειες. Θέλουμε να μειώσουμε το επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες, η νανοτεχνολογία, η κλωνοποίηση. Οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν αυτά τα πράγματα και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει μια κοινοτική ρύθμιση πώς θα διαμορφώνεται η πληροφόρηση, η ενημέρωση των καταναλωτών και ποιοτικά και ποσοτικά. Θα πρέπει οι εταιρείε που παράγουν τρόφιμα να υπομισθούν αυτέ τι ευθύνε. Γι' αυτό ο κανονισμό για τα τρόφιμα έχει τεράστια σημασία για την Ουγγρική Προεδρία, αυτό το νέο πλαίσιο. Πέρα από αυτά υπάρχει μια τροποποίηση τώρα για την οδηγία και για τους χυμούς, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις νέες αυτές ανάγκες των καταναλωτών στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε. Μέσα σε αυτή την τροποποιημένη οδηγία υπάρχουν νέα στοιχεία. Οι νέες ε, διατάξεις διαφοροποιούν μεταξύ χυμού και χυμού από συμπυκνωμένη ε, ουσία, από, από συμπύκνωση ε, φρούτων. Υπάρχουν και τα θέματα της ε, χρήσης γευστικών ουσιών και τώρα ε, οι ντομάτες εντάσσονται στον ε, κατάλογο των φρούτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φρουτοχυμών. Και τώρα Κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στο μέλλον δεν θα μπορεί η ε, ζάχαρη να αναμειγνύεται με φρουτοχυμούς. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται ζάχαρη σε φρουτοχυμούς. Στο μέλλον φρουτοχυμή θα είναι φρουτοχυμή και δεν θα προστίθεται, δεν προστίθεται σε αυτούς ζάχαρη. Όσο αφορά τη χρήση νέων τροφίμων, αυτή η πρόταση έχει ήδη υποβληθεί υπάρχει από το 2008 αλλά στην, ούτε και σε πρώτη ούτε και σε δεύτερη ανάγνωση μπόρεσε να επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Το Συμβούλιο τον Αύγουστο 2010 ξεκίνησε με τη δεύτερη ανάγνωση. Η Βελγική Προεδρία είχε τρεις φορές ήδη άτυπους τριμερείς διαλόγους ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Αυτή η συνδιαλλαγή ξεκίνησε επίσημα, αυτή η διαδικασία συνδιαλλαγής, ε, στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Το Συμβούλιο τι έκανε. Αυτά τα οποία ενέκρινε ως Κοινοβούλιο συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση δεν τα ενέκρινε. Και σαν συνέπεια αυτού, αυτής της απόρριψης, πρέπει τώρα η Επιτροπή Συνδιαλλαγή, συνδιαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 224 μέσα σε προθεσμία 6 εβδομάδων να επανασυγκληθεί, να επαναλειτουργήσει δηλαδή η διαδικασία συνδιαλλαγής. Η Ουγγρική Προεδρία τώρα στη συνέχεια ήδη στις 18 Ιανουαρίου 2011 ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα. Και αυτό που έκανε ήταν, υπήρξε κάποια πρόοδος όσον αφορά το, ε, την ε, εκτέλεση. Δεν είναι όμως ε, απλή η σημείο, να, δεν είναι απλό να σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με τα κλωνοποιημένα ε, ζώα και οργανισμούς. Εδώ πρέπει να γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσεις για να σημειωθεί πρόοδος. Είμαστε πρόθυμοι να διαβουλευτούμε και να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε αυτός ο κανονισμός το δυνατόν πιο γοργά να μπορέσει να εγκριθεί. Και από αυτού θα επανέλθω στη συνέχεια στην απάντηση ε, ερωτήσεων υστερότερα. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με τα τρόφιμα που θα διατίθενται στους καταναλωτές είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Η πληροφόρηση, οι αναφορές προς τους καταναλωτές στη συσκευασία για τα τρόφιμα. Όταν θα εγκριθεί αυτός ο κανονισμός θα ε, επικαιροποιηθεί και το θέμα τη της ετικετοποίησης στη συσκευασία. Ένα υποχρεωτικό στοιχείο για παράδειγμα που πρέπει να αναφέρει την πρόσθετη αξία που προσφέρει ένα τρόφιμο. Α, να είμαστε έτσι να αντιστοιχούμε αντιστοιχίσουμε το πιο αυστηρό πλαίσιο για τις ετικέτες και την τις ενδείξεις στις ετικέτες ώστε να συνειδητοποιούν πιο εύκολα και άμεσα οι αγοραστές, οι καταναλωτές τι προϊόν αγοράζουν και τι τους προσφέρει ακριβώς αυτό το προϊόν ως πρόσθετη αξία. Υπάρχει μια πολιτική συμφωνία και σε πρώτη ανάγνωση ε, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι το Φεβρουάριο θα εγκριθεί η πρόταση. Έτσι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ε, η Ουγγρική Προεδρία σε δεύτερη ανάγνωση με το Ευρωκοινοβούλιο επ' αυτών των θεμάτων. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη καρποφόρα συνεργασία με την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή. Και κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, τούτων λεχθέντων τώρα θα ήθελα να περάσω και να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Υπήρξαν αρκετές αίτιε ερωτήσεις. Ε, νέου είδου τρόφιμα, novel food, κλωνοποίηση ζώων ήταν ένα άλλο θέμα. Για παράδειγμα, εν μέρη μπορώ να πω ότι Ήδη είχα, προαναφέρθηκα σε κάποια στοιχεία. Ήδη προανέφερα για παράδειγμα για, στην Επιτροπή ε, Συνδιαλλαγής ε, πιο πριν. Όσον αφορά τώρα τα νέα τρόφιμα, food, σε σχέση με κλωνοποιημένα ζώα και την ε, τους απογόνους ε, των ε, ε, κλωνοποιημένων ζώων. Αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που έχει μεγάλη σπουδαιότητα και πρέπει να στρέψουμε σε αυτό το βλέμμα με ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη τώρα υπάρχουν διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο επίπεδο κορεπέρ στο επίπεδο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, πρέσβεων δηλαδή. Μετά έχουμε και θέματα σε σχέση με τη διοξίνη, ερωτήσεις που μου διατυπώθηκαν. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά τόσο τους καταναλωτές ε, αλλά εξίσου από την άλλη πλευρά και τις μονάδες ε, που ασχολούνται με την ε, που, κτηνοτροφικές μονάδες. Πρέπει να λάβουμε μέτρα που θα οδηγήσουν στο να αποφευθούν τέτοιου είδους σκάνδαλα στο μέλλον. Σκανδαλώδεις υποθέσεις όπως η μόλυνση με τις διοξίνες που σημειώθηκε με τα λύπη στην Γερμανία. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα σε τέτοιες κτηνοτροφικές ε, ε, μονάδες που θα διασφαλίζει, θα ε, κατοχυρώνει την ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία έχουν προταθεί από την Γερμανία και έχουν ξεκινήσει είναι ασφαλή μέτρα. Η συνεργασία όσον αφορά και την εποπτεία σε θέματα, τα κτηνιατρικά θέματα πρέπει να είναι λειτουργική. Και όντας λειτουργική είναι έχει ιδιαίτερη ε, σπουδαιότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σαν αυτή την μόλυνση ε, από διοξίνες. Ο Επίτροπος Ντάλι την Δευτέρα υπέβαλε μία πρόταση προς το Συμβούλιο στην οποία προβλέπεται, σύμφωνα με την οποία θα πρόκειται για θέματα αδειοδότησης ε, νέων μονάδων και για την αδειοδότηση σε σχέση με παραγωγούς τροφίμων όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης θα διέπονται από ένα πιο αυστηρό ε, πλαίσιο. Θα διαφοροποιούνται οι κατηγορίες πλέον ε, παραγωγής. Δεν θα συνδέονται ή δεν θα υπάρχει σύγχυση σε σχέση με την παραγωγή λοιπόν ή άλλων ουσιών. Θα πρέπει ένα νέο σύστημα monitoring, εποπτείας να δημιουργηθεί, ένα νέο σύστημα ε, τράπεζας δεδομένων, μια νέα τράπεζα δεδομένων, υποχρεωτική αναφορά άμεσα θα πρέπει να γίνεται για τέτοιου είδους ε, γεγονότα όταν θα υπάρχει κάποιο έβριμα θετικού χαρακτήρα, κάποια ανείχνευση ε, η οποία θα αποβαίνει θετική. Όλα αυτά είναι αναγκαία μέτρα που πρέπει στο μέλλον να βοηθήσουν ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδου σκάνδαλα σαν αυτό τη διοξίνη όσον αφορά τρίτε χώρε και την εισαγωγή και σεβασμό αυτών των ρητρών, όσον αφορά την μέτρηση, τον τρόπο μέτρηση ε, και τις διεργασίε. Όλα αυτά δημιουργούν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Εμείς εισάγουμε πολλά προϊόντα από τρίτες χώρες. Πρέπει να απαιτούμε να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές και ρήτρες έναντι αυτών των προϊόντων από τρίτες χώρες που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιες προδιαγραφές και συνθήκες παραγωγής πρέπει να ισχύουν για αυτά τα προϊόντα κατά την παραγωγή τους από τρίτες χώρες, μια και εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν αυτά τα προϊόντα, σαν αυτές οι συνθήκες και ρήτρε που ισχύουν για την παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέθηκαν κάποια άλλα ερωτήματα εξάλλου για τα τρόπο, τα γενετικά τροπο, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους για αυτό το ζήτημα. Και φυσικά και οι πολίτες είναι διχασμένοι, έχουν διαφορετικές απόψεις. Ενδιαφέρονται όμως πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια δέσμη μέτρων για τα γενετικά τροποποιημένα και από πλευράς των κρατών μελών δίνεται πλέον μεγαλύτερη ελευθερία να προβούν σε ρυθμίσει τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αν κάποια κράτη-μέλη επιθυμούν στην επικράτειά του να προβούν στην έγκριση και αδειοδότηση καλλιεργειών γενετικά τροποποιημένων φυτών και οργανισμών ή όχι. Αυτό έχει ένα θετικό μήνυμα το οποίο συνεπάγεται, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τι επιφυλάξει και τι ενστάσει των κρατών μελών και προσπάθησε να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα με αυτή την πρόταση. Η Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει να επιτηρεί ε, την κατάσταση και θα θεωρεί και θα δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στον κανονισμό για τα γενετικά τροποποιημένα. Η νομοθετική πρόταση σε σχέση με αυτό το ζήτημα ε, συνάδει και ανταποκρίνεται με την πρόταση του κυρίου Μπαρόζο. Ο κύριος Μπαρόζο στο πρόγραμμα εργασίας του που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εντάξει αυτό το θέμα και συμφώνησε το Ευρωκοινοβούλιο τότε με αυτή την ε, αντιμετώπιση. Θεωρώ εξίσου σημαντικό να αναφέρω εξάλλου ότι ίσως για την ασφάλεια ένα σύστημα ρητρών ή δικλείδων ασφάλειας δεν θα αλλάξει, θα παραμείνει αναλύωτο και έτσι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να είναι σε θέση από πλευρά τους ε, να κάνουν λόγο, να ρυθμίζουν αυτές τις ρήτρες ασφάλειας ε, ε, όπως ε, επιθυμούν σε σχέση με το πλαίσιο ρύθμισης που θα ισχύει στην επικράτειά τους για τα γενετικά τροποποιημένα, την έγκρισή τους ή την απαγόρευσή τους και σε ποιο εύρος θα επιτρέπεται να καλλιεργούνται κτλ. κτλ υπόψη κοινωνικά, οικονομικά και άλλα επιχειρήματα. Προσπαθούμε όμως τώρα να καταλήξουμε σε μια εναρμονισμένη κοινή λύση που θα ισχύει σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την ΕΦΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια ασφάλεια τροφίμων. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής είναι η υπηρεσία ακριβώς για την ασφάλεια των τροφίμων και έχει ένα δρομολόγιο, ας το πω έτσι, οδηγίες ε, που έχει συντάξει για την αξιολόγηση κινδύνων. Θα επανεξεταστεί αυτή η όλη προσέγγιση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναθεώρηση όμως αυτή. Και έτσι είμαι πεισμένος πρέπει να πω μέσα στο πλαίσιο αυτό ότι οι ανεξάρτητοι επαΐοντες, οι ανεξάρτητοι ετησία όσον αφορά στην, στον απολογισμό και στην εκτίμηση των επιπτώσεων είναι πολύ μεγάλη σημασία θέμα. Πρέπει να υπάρχει αντικειμενική, ανεξάρτητη ε, δυνατότητα αξιολόγηση. Το βλέπουμε αυτό και σε σχέση και με την αδειοδότηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι επιχειρήσεις πρέπει δειγματοληπτικά να υποβάλουν ε, δειγματοληπτικά ε, κάποια στοιχεία. Αυτά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, αυτοί οι έλεγχοι δεν έχουν μπορέσει ακόμα να ολοκληρωθούν. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, τέτοιες προβληματικές καταστάσεις και να ε, βρούμε λύσεις. Εν τέλει, η ετικετοποίηση των τροφίμων είναι και αυτό ένα θέμα. Θα ήθελα να σας εκφράσω κάποιες σκέψεις μου για αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο για απομιμήσεις ή για υποκατάστατες ουσίες, ουσίες υποκατάστατα έχει ήδη προβεί σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η θέση του Συμβουλίου συνάδει με τις ε, τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βέβαια. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να ενημερώνουμε καλύτερα τους καταναλωτές σε σχέση με την ε, ε, συμπερίληψη τέτοιων ουσιών ή όχι. Έχουμε ένταξη λοιπόν αρχών και κατευθυντήριων, ας το πω έτσι, αρχών σύμφωνα με τις οποίες οι περιπτώσεις παραπλάνησης θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. Διότι στα τρόφιμα πρέπει πάντα να αναφέρεται όταν και αν εμπεριέχονται παραδοσιακές, ε, παραδοσιακές ουσίες για την παραγωγή ενός, ενός τροφίμου ή υποκατάστατα ως ουσίες. Αν καταλήξουμε σε αυτή την προσέγγιση τότε σε αυτή τη διαφοροποίηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραδοσιακή ονομασία μιας ουσίας στην παρασκευή ενός προϊόντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν το όνομα μιας παραδοσιακής ουσίας όταν έχει υποκατασταθεί από υποκατάστατο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τρεις ερωτήσεις για σας. Αρχίζουμε από την κυρία Λιωτάρ Κυρία Ροτμπάρεν, θέλετε και εσείς να παρέμβετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι θα είναι πιο χρήσιμο να συνεχίσουμε σε διμερές επίπεδο και όχι στο πλαίσιο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ja, Καλώς, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και για την εισαγωγική σας παρέμβαση. Και ε, ιδιαίτερα δε και για την παρουσίαση για την ασφάλεια των τροφίμων. Εγώ είμαι η συγγήτρια για τα καινοτόμα τρόφιμα, novel foods, όπου ε, πρόκειται να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία συνδιαλλαγής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για τις προσπάθειες που κατέβαλε ήδη από τις πρώτες ημέρες της Προεδρίας για την υποβολή ενός εγγράφου. Και αυτό πραγματικά είναι ευχάριστο. Όπως ήδη ελέγχθη εδώ, τα καινοτόμα τρόφιμα, ουσιαστικά είναι τρόφιμα τα οποία παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα και 77% ε, των ε, πολιτών της Ευρώπης δεν θέλουν τέτοια προϊόντα και κατά τη δεύτερη ανάγνωση η θέση του Κοινοβουλίου ήταν απολύτως σαφής. Ελέγχθη ότι ε, τα τρόφιμα τα οποία προκύπτουν από, το, από ζώα δεν θα πρέπει να περιληφθούν τον κατάλογο αυτό των καινοτόμων τροφίμων. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Τώρα λοιπόν η Κομισιόν μας λέει ότι θα έρθει με μια δεύτερη ε, πρόταση που συνδέεται με την κλωνοποίηση. Πρέπει λοιπόν να ανεβρεθεί μια λύση. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί. Εγώ λοιπόν προτείνω το που θα προταθεί να είναι νομικά δεσμευτικό, ώστε ε, να αποφύγουμε στο μέλλον να υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς Κομισιόν προς άλλη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε τρόφιμα από κλωνομημένα προϊόντα και δεν θα πρέπει να κυκλοφορήσουν αυτά ε, στην αγορά. Πρέπει λοιπόν η νέα νομοθεσία να περιλαμβάνει συγκεκριμένο άρθρο ε, ώστε όλη η ισχύουσα νομοθεσία να ε, θεωρηθεί απειρχαιωμένη όταν θα εισαχθεί η νέα νομοθεσία. Εικάζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση ή μια κοινή δήλωση εξ των τριών θεσμικών οργάνων με, με, με, στόχο να λέει ότι ε, αυτού του είδους τρόφιμα δεν είναι εγκεκριμένα, δεν έχουν άδεια. Δεν θα δίδεται άδεια στα τρόφιμα αυτά. Και δεν θα έχουν καμία δυνατότητα επιτυχίας του στόχου τους αν ε, καταφύγουν στα δικαστήρια. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορεί να προσφέρει η Ουγγρική Προεδρία ως λύση. λύση με την οποία θα συμφωνήσουν τόσο Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο. Να είναι όμως μια νομικά δεσμευτική λύση εν ώψη της νέας νομοθεσίας ε, για την κλωνοποίηση. Δεύτερον, ε, είπατε ότι έχει σημειωθεί προόδος και στις ενέργειες όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων. Σημαίνει ότι το Συμβούλιο έχει λάβει τελική οριστική απόφαση από αυτού. Έχω μία ερώτηση σχετικά με το περιβάλλον. Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν μπορώ να υποβάλω την ερώτηση. Ναι, ωραία, προχωρήστε, παρακαλώ. Είμαστε μέλη του Κοινοβουλίου, όλα είναι εφικτά. Η Ουγγρική Προεδρία έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη. και η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από εσά. Η φήμη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ε, και αφορά την νομοθεσία και την ε, εφαρμογή της στις χώρες μέλη. Ε, έγινε μάλιστα σχετικό σχόλιο από την κυρία Χάσα σήμερα το πρωί. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για ποιο λόγο η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την ε, κόκκινη λάσπη πήρε άδεια, μάλλον παράταση της άδειας λειτουργίας της μέχρι το 2018. Και δεύτερον, μπορείτε να ε, μας διαβεβαιώσετε ότι θα υπάρξει μεταφορά νέας τεχνολογίας στους προσεχείς 6 μήνες και αυτή τη μεταστροφή της τεχνολογίας το κόστος ποιος θα το πληρώσει. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε για το γεγονός ότι η κυρία Ροτ Μπέρεντ αποχώρησε ήδη. Κάπως με εξέπληξε αυτό για το ότι ε, ανέφερε κάποια πράγματα και τώρα αποχώρησε. Τώρα δεν πρέπει ούτε τον κύριο Λάινεν ούτε τον κύριο Φαζέκα να υπερασπιστώ. Εντάξει, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι στην ημερήσια διάταξη είχε εξειδικευθεί ότι θα υπήρχαν δύο ακροάσεις. Ότι θα υπήρχε η δυνατότητα ο κύριος Φαζέκας επί δύο θεμάτων να τοποθετηθεί δεν γίνεται ο κύριος Λάινεν ή ο κύριος ε, Φαζέκας ε, για την ασφάλεια των τροφίμων να μην κάνουν καθόλου λόγο και σε αντίθεση με όλα αυτά επρόκειτο για το γεγονός ότι ο κύριος Φαζέκας για μια πολύ ιδιαίτερη προτεραιότητα ήθελε έπρεπε να τοποθετηθεί και γι' αυτό εξεφώνησε και ξεχωριστή παρέμβαση επ' αυτού του θέματος. Τώρα όσον αφορά τη διοξίνη σε σχέση με τις διοξίνες την Δευτέρα ήδη ασχοληθήκαμε διεξοδικά με το θέμα. Δεν θέλω τώρα να υπησέθουμε περισσότερο σε αυτό. Θα ήθελα όμως περισσότερο κάτι άλλο να κάνω. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός ήδη την Δευτέρα κατέληξε σε μια συμφωνία, μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία και βλέπουμε τώρα το φως στο τέλος στη σύραγγα, ε, στην άκρη του τούνελ. Βλέπουμε λοιπόν ε, τι μπορεί να γίνει. Ετέθη μια ερώτηση και λέμε καμιά φορά στην Ουγγαρία σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε η Ουγγαρία να μην γίνει η χωματερή τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα είδος χωματερής για τα τρόφιμα της υπόλοιπης Ευρώπης πρέπει να καταβάλει όμως προσπάθειες η, Ευρώπη, η Ευρώπη ώστε να μην γίνει η Ευρώπη χωματερή τροφίμων του υπόλοιπου πλανήτη. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τα προϊόντα, τα τρόφιμα από τρίτες χώρες, από την αλλοδαπή δηλαδή, από το εξωτερικό, υπό ακριβώς τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις να παράγονται όπως τα τρόφιμα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει η εποπτεία, να, η αναγκαία επιτήρηση, να γίνονται έλεγχοι, να υπάρχουν αυστηρότατες κυρώσεις και θα πρέπει τα μολυσμένα τρόφιμα να παραμένουν εκτός Ευρώπης οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα αμέσω να δώσω συνέχεια όσον αφορά τους προλαλήσαντες και θα ήθελα συγκεκριμένα να τοποθετηθώ σε αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν από τον κύριο Άντα. Υπέ, ε, υπέβαλα μια γραπτή ερώτηση προς τον κύριο Νταλή, εγώ ο ίδιος, που αναφερόταν στο εξή. Γιατί έλεγα, έλεγε η ευρωπαϊκή νομοθεσία καθιστά εφικτό σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων διασυνοριακά, στην εισαγωγή τροφίμων να συμβαίνουν, να έχουμε δύο μέτρα και σταθμά σε σχέση με τα εντό παραγόμενα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παραγόμενα εκτό που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα εισαγόμενα τρόφιμα, τέτοιου είδου, για παράδειγμα, ουσίε μπορούν να χρησιμοποιούνται όπω αυτέ που απαγορεύονται ήδη προπολού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι έργο του ε, Συμβουλίου, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο είτε να πείσει τον κύριο Ντάλι το γεγον, για το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή διαφορετικά το Συμβούλιο να μπορέσει να ε, καταλήξει σε μια δήλωση, σε μια διακήρυξη λέγοντας το ίδιο ότι αυτό το πλαίσιο νομικό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Θέλετε να κλείσετε παρακαλώ τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, Πρόεδρε. Και σε σχέση με το σκάνδαλο των διοξινών, φυσικά ασχολούμεθα και μας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος το γεγονός ότι η Ουγγρική Προεδρία ήδη κατά την πρώτη της συνεδρίαση ήδη μπόρεσε να πετύχει ένα, μια κοινή θέση από πλευρά των κρατών μελών στο Συμβούλιο και για την λήψη μέτρων όπως εξέθεσε σχετικά τα θέματα αυτά ο κύριος Νταλή. Και τώρα κάτι άλλο. Πιστεύω ότι η αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε οδήγησε σε αυτή την επιτυχία. Τίποτα άλλο δεν ήταν παρά αποτέλεσμα επιτυχούς συνεργασίας. Μπορεί ουσίες σε τρίτες χώρες να αδειοδοτούνται και να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και έτσι να διοχετεύονται στην αγορά τρόφιμα που εμπεριέχουν τέτοιες ουσίες. Αυτές όμως οι ουσίες απαγορεύονται, να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτό είναι δεδομένο και συμβαίνει. Έχουμε διαφορετική ορους όρους και προϋποθέσεις. Και λόγω των συμφωνιών του ε, Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Αν τέτοιου είδους ουσίες και προϊόντα δεν συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία. Και η ΕΦΣΑ, η Οργανισμός η Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ελέγχει αυτά τα τρόφιμα. Πέρα από αυτό υπάρχουν οριακές τιμές οι οποίες ε, ισχύουν και έχουν εγκριθεί και εντάσσονται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε όμως μόνο λαμβάνονται υπόψη, τότε μόνο ε, μπορεί να εισαχθεί ένα τρόφιμο και ε, όταν δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από όλα αυτά απορρέει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και υπόσχομαι ότι κατά την επόμενη συνάντησή μου μαζί του θα συζητήσω το θέμα με τον κύριο Νταλή. Τώρα όσον αφορά την ε, περίπτωση κόκκινης λάσπης αυτής της ε, ε καταστροφής στην ε, Ουγγαρία θα πρέπει πιο εξειδικευμένα να συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί υπόψη και η εσωτερική κατάσταση των πραγμάτων από πλευρά νομοθεσία στην Ουγγαρία. Υπήρχε ένα κυβερνητικό κανονισμό του 1996 στην Ουγγαρία που την Ερυθρά Λάσπη την ε, αξιολογούσε ω ε, επικίνδυνο απόβλητο. Το 2002 η τότε, το τότε Υπουργείο ε, Προστασίας του το τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο του εναρμονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κάποιες, ε, ε, κάποια νέα πλαίσια και επικαιροποίησε αυτο τον κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία πλέον υιοθετήθηκε και τα πράγματα άλλαξαν. Έτσι, ένας υπουργικός κανονισμός υιοθετήθηκε ο κανονισμός 2001 κάθετος 16 που καθιστούσε ε, δυνατό να ε, θεωρείται απόβλητο ε, η ερυθρά λάσπη που ήταν υποπροϊόν της παραγωγής αλουμινίου και έτσι είχαμε και την εγγραφή, την ένταξη ουσιών στον κατάλογο επικινδύνων αποβλήτων. Η νέα αυτή ο νέος αυτός ουγγρικός ε, κανονισμός ε, άρχισε να ισχύει το 2002 και καθόριζε ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο παραγωγός ε, του εκάστοτε, της εκάστοτε ουσίας ως, αποβλη, ως αποβλήτου είναι εκείνος μπορούσε να αποφασίζει αν η ερυθρά λάσπη θα ίσχυε, θα εντασσόταν στα επικίνδυνα απόβλητα ή όχι. Αυτή ήταν η κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Ουγγαρία μετά από αυτά τα νομοθετήματα. Η επιμέρους τώρα αυτή η μονάδα παραγωγής, αυτή η βιομηχανία ήδη στις 19 Δεκεμβρίου 2001 είχε ενημερώσει τις αρμόδιες ουγγρικές αρχές για το γεγονός ότι η ερυθρά λάσπη μελλοντικά θα δεν θα θεωρεί το επικίνδυνο απόβλητο ως υποπροϊόν της ε, διαδικασίας παραγωγής αλουμινίου από αυτή την βιομηχανία. Η αρμόδια λοιπόν Ουγγρική Αρχή ενέκρινε το αίτημα να μην είναι επικίνδυνο απόβλητο και μετά από το 2002 Εφ' εξής, υπήρξε ενημέρωση ε, ότι θα πρέπει δειγματοληπτικά μέσα από δειγματοληπτικούς ελέγχους να αποδεικνύει η βιομηχανία αυτή ότι πραγματικά η ερυθρά λάσπη δεν, ήταν, δεν θα ήταν επικίνδυνο απόβλητο. Εδώ υπήρξαν ε, λοιπόν επιστημονικές αναλύσεις και εξετάσεις που καταδείκνυαν, αποδείκνυαν ότι δεν ήταν επικίνδυνη λάσπη αυτό το, ε, δεν ήταν επικίνδυνο απόβλητο αυτή η ερυθρά λάσπη. Έτσι καταλήξαμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ε, αποφάνθηκε αυτή λέγοντας ότι η ερυθρά λάσπη ανταποκρινόταν στις νομικές διατάξεις που ίσιαν και που εντασσόταν έτσι η ερυθρά λάσπη στην κατηγορία μη επικίνδυνων αποβλήτων. Τελεία και παύλα. Αυτή η ερυθρά λάσπη λοιπόν ε, εντάχθηκε στην κατηγορία των διασπόμενων ε, ουσιών ή αποβλήτων και δεν εντάχθηκε ως τοξικό απόβλητο στον αντίστοιχο κατάλογο. Η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Σεπτεμβρίου 2011 άσκησε επικρίσεις λέγοντας ότι οι Ουγγρικές αρχές δεν τήρησαν με σωστό τρόπο τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές η Ουγγαρία μετά από αυτές τις επικρίσεις ε, ενέκρινε ένα νομοθέτημα το οποίο είναι το νομοθέτημα 2010-181 το οποίο ανέφερε ότι η ερυθρά λάσπη που σε σχέση με την παραγωγή βοξίτη, επεξεργασία βοξίτη είναι υποπροϊόν, επικίνδυνο υποπροϊόν, επικίνδυνο απόβλητο. Και γι' αυτό οι νομικές διατάξεις ε, θα πρέπει να ισχύουν όπως ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα σε σχέση με την παραγωγή ερυθράς λάσπης. Από τότε δόθηκε λοιπόν εντολή στις αρμόδιες εποπτικές αρχές να ασκήσουν τους αναγκαίους ελέγχους σε σχέση με αυτή τη μονάδα. Αυτή είναι σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με το παρόν η προηγούμενη και η παρούσα νομική βάση και το νομικό πλαίσιο. Τώρα χρησιμοποιείται μια νέα τεχνολογία στεγνής ή ξηρής παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ως υποπροϊόν η δημιουργία ερυθράς λάσπης κατά την παραγωγή αλουμινίου. Και τώρα έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, δεν έχουμε ως ε, υποπροϊόν κατά τη διάρκεια των ε, διαδικασιών παραγωγής έρυθρα λάσπη πλέον. Είμαστε πεισμένοι ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες από πλευρά μας όπως έπρεπε. Το θεώρησα σημαντικό να επισέλθω σε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς έχει το σημερινό νομικό καθεστώς, ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ή πώς τροποποιήθηκαν οι τεχνολογίες κατά την παραγωγή αλουμινίου. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο πλέον και όσον αφορά το θέμα της κλωνοποίησης, η Προεδρία του Συμβουλίου έχει συνειδητοποιήσει απόλυτα πόσο επίμαχο είναι αυτό το θέμα και ότι οι πολίτες θεωρούν ότι δεν επιθυμούν να καταναλώνουν ε, κλωνοποιημένα ε, ζώα στα προϊόντα που αγοράζουν και είμαι βέβαιος ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση και συμφωνία. Ίσως θα πρέπει να υπάρξουν ευρύτερες διαπραγματεύσεις βέβαια και διαβουλεύσεις για να επιτευχθεί αυτό ως αποτέλεσμα. Υπάρχει εδώ όμως ε, από πλευράς της Προεδρίας του Συμβουλίου με την έγκριση των τριών μεγάλων θεσμικών οργάνων η δυνατότητα να προβούμε σε μια τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε από τη σημερινή συζήτηση ότι η στοχοθέτησή μας και για την ασφάλεια τροφίμων αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος οι στοχοθετήσεις μας είναι κοινέ και ενιαίες. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, να υπηρετήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και να μπορέσουμε να πετύχουμε να ζούμε σε ένα πλαίσιο αξιοπρεπές για τους τους Ευρωπαίους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της υγείας και της, υπεράσπι... της προστασίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υγείας των πολιτών. Και οι στόχοι του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας προς αυτό στοχεύουν. Θέλουμε η πολυμορφία στη γεωργία μας να διασφαλιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε μας κάνατε την τιμή να είστε μαζί μας σήμερα το πρωί και που απαντήσατε ε, με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο στις ερωτήσεις που ετέθεσαν από τους συναδέλφους και νομίζω ότι ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμες και επικοδημητικές. Σας ευχαριστώ θερμά.